Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ πολύ καθίστε για να ξεκινήσουμε άμεσα με τις εργασίες μας. Έχουμε πολλά σημεία να καλύψουμε στη μερίσια διάταξη. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις εργασίες μας και Πάμε στο σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης. Κανονικά προβλεπόταν για χθε το απόγευμα, δεν καταφέραμε να το καλύψουμε για πρακτικούς οργανωτικούς λόγους και αναφέρομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεολαία. Θα ήθελα ευθύ αμέσω να δώσω τον ε, λόγο στην εισηγητή μας, τον κύριο Ματέο Μπιάνκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα το ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω την γνωμοδότησή μου, η οποία ομόφωνα εγκρίθηκε στην Επιτροπή ΣΕΝΤΕΚΑ. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε και εδώ με μεγάλη πλειοψηφία να καταφέρουμε να υπερψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Δεν έχω λάβει τροπολογίε. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου για την υποστήριξη που έδειξαν προ την γνωμοδότηση αυτή. Τη γνωμοδότηση αυτή τη συντάξαμε μετά από πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Σώματο Αλληλεγγύη και για μια νέα στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την νεολαία. Η γνωμοδότηση αυτή ουσιαστικά έχει μια έντονα τοπική και περιφερειακή διάσταση. Πιο συγκεκριμένα, ήθελα στη γνωμοδότηση αυτή να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σώματο Αλληλεγγύη και γενικά στα προγράμματα τα θελοντικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να συμμετέχει περισσότερο η περιφερειακή και η τοπική διάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εντάξουμε τα ήδη φυστάμενα προγράμματα στο τοπικό επίπεδο όσον αφορά την εθελοντική συμμετοχή των νέων. Ήρθα σε επαφή επίση και με τον αρμόδιο εισηγητή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από κοινού είπαμε ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Η γνωμοδότηση, λοιπόν αυτή τονίζει ότι θα πρέπει να τονιστεί το τοπικό επίπεδο. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που σε τοπικό επίπεδο συμμετέχουν σε θελούσια προγράμματα τα οποία θα πρέπει να ενσωματωθούν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη. Είναι προγράμματα τα οποία βοηθούν πάρα πολύ και το αστικό θεματολόγιο αλλά και τη διαχείριση τη ε, μεταναστευτική ροή. Ανταποκριμόμενη επίση στη νέα στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την νεολαία, η γνωμοδότηση αυτή τάσσεται υπέρ τη νέα αυτή στρατηγική και χαίρεται πάρα πολύ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διορίσει έναν συντονιστή για τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεολαία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε εδώ πέρα μία εκπεριτροπής, ένα εκπεριτροπή συντονισμό ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και τον EU Youth Coordinator. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να καλύψουμε όλε τι κοινωνικέ απαιτήσει σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο όσον αφορά την πολιτική για του νέου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να σωματώσουμε τη διάσταση των νέων σε όλε τι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο οι θύνοντε σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο τόσο από το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε πραγματικά να ανταποκριθούμε στι κοινωνικέ ανάγκε των νέων σε τοπικό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να έχουμε μια αυθεντική συμβολή των νέων οι οποίοι θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στα κοινά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο διαρθρωμένο λοιπόν διάλογο με του νέου θα πρέπει να εμπλέκει περισσότερο τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ. Είμαι πεπισμένο λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε και ένα σήμα ποιότητο όσον αφορά τα προγράμματα υπέρ των νέων. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε καλύτερη αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, καλύτερη συνεργασία και επίση καλύτερη συμμετοχή και των αθλητικών οργανώσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δείξουμε για όλα αυτά τα προγράμματα την απαιτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξη και ελεγγύη. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν παρατηρήσει στα πλαίσια τη γενική συζήτηση. Δεν βλέπω κανέναν. Μπορούμε τότε να περάσουμε ευθύ αμέσω τροπολογίε που, όπω ακούσαμε από τον εισηγητή, δεν έχουμε τροπολογίε. Άρα περνάμε ευθύ αμέσω στην τελική ψηφοφορία. Ποιο είναι υπέρ τη γνωμοδότηση, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Η γνωμοδότηση εγκρίνεται ομόφωνα. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια στον εισηγητή για όλη την εργασία του. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε έτσι στο σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης. Γνωμοδότης όσον αφορά τις γειτονικές χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο, εισηγητής εδώ πέρα είναι ο Hans Janssen. Κύριε Πρόεδρε και εσείς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι σύμπτωση που η γνωμοδότησή μου σχετικά με τις γειτονικές χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο συζητείται σήμερα, όπου σήμερα συζητείται και το Brexit η Βρετανική αποχώρηση και θα τοποθετηθεί αργότερα ίδιος ο κύριος Μπαρνιέ για το θέμα αυτό. Δεν είναι άλλωστε σύμπτωση που σύντομα θα θεωρούμε γειτονική χώρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Το δε Brexit σιγά σιγά μάλιστα βλέπουμε να αναπτύσσεται το αίσθημα ότι ίσως ορισμένοι μετανιώνουν και ίσω επιτέλους, ε, δηλαδή, μάλλον αργότερα, το Ηνωμένο Βασίλειο να επανέλθει ω υποψήφια προς ένταξη χώρα. Εν πάση περιπτώσει βρίσκω ότι το θέμα ταιριάζει στη σημερινή ημέρα. Πρέπει να εξετάζουμε τι συμβαίνει και εκτός Ευρωπαϊκής Υπήρου. Γιατί ούτω ή άλλω εδώ έχουμε αρκετά θέματα εμεί να συζητήσουμε. Ο πατέρας μου που είναι 88 ετών λέει συχνά ότι έξω από την πόρτα σου υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Local is global και το ανάποδο. Μιλώ για τις γειτονικέ μας γεωγραφικά χώρες. Είναι πραγματικά γείτονες ή είναι γείτονες άλλων. Έχουμε και εμείς μια ευθύνη για τις χώρες αυτές και για την παγκόσμια πολιτική. Πρόκειται και για τις ε, γειτονικέ χώρες σε γειτονικές υπήρους επίσης. Και εάν η κοινωνική και οικονομική τους ανάπτυξη είναι θετική για τους πολίτες τους ή εάν οδηγεί εν τέλει τους πολίτες αυτούς να έρθουν να χτυπούν τη δική μας πόρτα επειδή θεωρούν ότι εδώ θα περάσουν καλύτερα. Άρα, ήδη το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Το ερώτημα είναι τώρα για εμάς ως Επιτροπή Περιφερειών. Εάν οι οργανισμοί μας τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης με τα 123 δισεκατομμύρια ευρώ του κοινοτικού προϋπολογισμού αν εξυπηρετούνται επαρκώς, αν συμφωνούν. Αν αρκούν δηλαδή τα κονδύλια αυτά για να μπορούμε να παίξουμε σωστά το ρόλο μας και εμείς ως οργανισμοί τοπικής και περιφερικής, και περιφερικής αυτοδιοίκησης. Γιατί έχουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ για να φροντίσουμε τις σχέσεις μας με άλλες γειτονικέ περιφέρειες. Και οι ευρωβουλευτές έχουν δεχθεί την ιδέα αυτή και γι' αυτό έχουν προβλέψει σχετικά στις εκθέσεις τους. Έχουμε και τροπολογίες οι οποίες ελπίζω να ε, υπερχιστούν εδώ και να βρουν και απήχηση και στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, θέλω να μιλήσω για την ουδέτερη στάση απέναντι το σύμφωνο για τη μετανάστευση των Ηνωμένων Εθνών. Γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση και πώ διαμορφώνεται η πολιτική κατάσταση γύρω από το θέμα αυτό στο Βέλγιο, για το Μαρακέσι δηλαδή. Θα δούμε τώρα πώ θα εξελιχθεί. Επίση θέλω να τονίσω του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών που πρέπει να του επαναλαμβάνουμε διαρκώ και να του έχουμε διαρκώ στο νου μα. Και τονίζω επίση ότι οι σημερινοί στόχοι των Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Ταμείων περιλαμβάνονται επίσης και πρέπει να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα κονδύλια. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους μου για, τις, ε, για τη συνεισφορά τους στην διαμόρφωσή της. Ευχαριστώ βεβαίως και τις συνεργάτηδες της Γραμματείας και την εμπειρογνώμονά μου, κυρία Τζέζι Πόστερ, η οποία εργάστηκε σκληρά για την σύνταξη της γνωμοδοτήσεως, η οποία γνωμοδότηση προέκυψε βέβαια από ομαδική εργασία και ελπίζω ότι έτσι θα βελτιώσουμε λίγο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Εισηγητά. Δεν βλέπω, λέει ο πρόεδρο. Α, με συγχωρείτε, Κάποιο είναι. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Γιάνσεν για την έκθεσή του. Νομίζω ότι το σχέδιο της, Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραβλέπει τις ε, τοπικές και περιφερειακές αυτοδιοικήσεις που συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη Υπάρχουν και πάρα πολύ θετικέ παραδόσει και στη Σουηδία και στι κάτω χώρε. Και η Γερμανία έχει αρχίσει τώρα να ενισχύει τον ρόλο των ε, τοπικών αυτοδιοικήσεων. Έχουμε συγκεκριμένε εμπειρίε και στην Παλαιστίνη και στην Ουκρανία, Μολδαβία, Τουρκία. Πρόκειται για έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ομοσπονδιακή Γερμανική Κυβέρνηση. Εάν τώρα υπάρξει ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σωστό και τονίζω επίσης ότι στον τομέα αυτό υπάρχει και μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη των περιφερειών. Δεν αναμένουμε ανταμοιβή, το κάνουμε και προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς το δικό μας. Και νομίζω ότι χρειάζεται μια συνολική χρηματοδότηση για αυτήν την διαπεριφερειακή συνεργασία και να ενισχυθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον ε, κύριο Συγητή. Εκφράζουμε ορισμένε επιφυλάξεις σχετικά με την αναφορά στο Παγκόσμιο ε, Σύμφωνο Μετανάστευσης. Υπάρχουν εκεί κάποια ασαφή σημεία και από τα οποία εκπηδούν κάποιες αμφιβολίες. Υπάρχουν και πλήρες χώρες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διατηρούν επιφυλάξεις ό,τι αφορά το Παγκόσμιο Σύμφωνο Μετανάστευσης. Και διαρωτώ με εάν είναι ορθό να το επισημαίνουμε σε τροπολογία την οποία έχει καταθέσει ο ίδιος ο εισηγητής. Δηλαδή στην τροπολογία αυτή αναφέρει το σύμφωνο αυτό και διαρωτώ με αν είναι πράγματι η κατάλληλη χρονική στιγμή. Η έκθεση κατά τα άλλα είναι εξαιρετική. Αλλά εάν θα πρέπει να μιλήσουμε σε αυτό το κείμενο εδώ για το Παγκόσμιο Σύμφωνο ε, Μετανάστευσης εμένα δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Έχω κάποιες επιφυλάξει. Ορίστε κύριε Κλεζό. Για να σχολιάσω αυτό που μόλις ελέγχθη. Στη Γαλλία διαμορφώνεται μια έντονη συζήτηση στα κοινωνικά μέσα σχετικά με το ότι το σύμφωνο της μετανάστευσης οδηγεί σε ξεπούλημα της Ευρώπης και της Γαλλίας και σε μια μετανάστευση χωρίς έλεγχο. Ο καθένα, νομίζω το υπενθυμίζει σήμερα και είναι σωστό να υπενθυμιστεί και εδώ, ότι το σύμφωνο αυτό είναι σύμφωνο συστάσεων. Δεν περιλαμβάνει νομικές δεσμεύσεις και σέβεται απολύτως την κυριαρχία των χωρών σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική πολιτική. Το βρίσκω λοιπόν δίκαιο να αναφέρουμε το σύμφωνο αυτό, το οποίο προσφέρει ένα ε, ανθρωπιστικό όραμα στη μετανάστευση και το οποίο ταυτόχρονα σέβεται την κυριαρχία των χωρών χωρίς να τους επιβάλλει πρόσθετες νομικέ δεσμεύσεις. Αντιθέτως λοιπόν εγώ υποστηρίζω την αναφορά που κάνει ο εισηγητή στο κείμενό του. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ορίστε παρακαλώ. Γιόγκμαν. Κύριε Πρόεδρε, και εμεί εξετάσαμε το κείμενο της ε, εισηγήσεω και την αναφορά στο Μαρακέσου και είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο ο εισηγητής αναφέρεται στην τροπολογία του στα γεγονότα μόνο. Για τη δική μας πολιτική ομάδα πάντως έχει καλός ο τρόπος με τον οποίο ε, μεταχειρίζεται το θέμα και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας και τις ευχαριστήσεις μας προς τον εισηγητή. Άλλος παρακαλώ, δεν βλέπω κανέναν άλλον να ζητεί να παρέμβει. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τι τροπολογίε. Τροπολογία 1 του εισηγητού, αντικατάσταση τη τροπολογία υπέρ, κατά, αποχέ. όχι ακόμη, δεν είπα ακόμη αποχέ ο πρόεδρος, με συγχωρείτε. Όχι, θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία. Όλες μαζί 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, α, αρκετές είναι μου φαίνεται. Αυτά τα, αυτές τις τροπολογίες λοιπόν όλε μαζί υπέρ, κατά, Αποχέ. δεν έχει αποχέ εγκρίθηκε. Τροπολογία 7 υπέρ κατά απορρίπτεται 8 που αντικαθιστά την αρχική 8 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 11 του εισηγητού υπέρ κατά εγκρίνεται Α, με, συγχωρείτε. Ναι, όχι, ε, δεν υπάρχει άλλη. Τελική ψηφοφορία επί της γνωμοδοτήσεως. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται η γνωμοδότηση με μία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά και σας ευχαριστώ για την ολοκληρωμένη αυτή εργασία. Και τώρα προχωρούμε στην γνωμοδότηση για το πρόγραμμα Invest EU, την οποία παρουσιάζει ο εισηγητής μας κύριος Αγοραστός. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Το InvestEU είναι ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο καλούμαστε να οικοδομήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση του μέλλοντος. Δεν είναι ένα απλό πρόγραμμα. Δεν αφορά μόνο τους οικονομολόγους, τους επιχειρηματίες, τα στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών. Το InvestEU αφορά κάθε Ευρωπαία και κάθε Ευρωπαίο. Αφορά τις νέες μητέρες που χρειάζονται παιδικούς σταθμούς και σχολεία για τα παιδιά τους. Αφορά τους νέους επιστήμονες που έχουν μια καινοτόμο ιδέα και θέλουν να την αξιοποιήσουν επιχειρηματικά. Αφορά τις εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται να εξασφαλιστούν πρόσβαση σε προσιτή χρηματοδότηση για να ανταπεξέλθουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αφορά τους ασθενείς που χρειάζονται και περιμένουν καινούριε θεραπείες. Αφορά στο τέλος τέλος όλους μας που θέλουμε και αξίζουμε να ζούμε σε ένα καθαρό περιβάλλον με σύγχρονες υποδομές. Θέλουμε να αξιοποιούμε τη δημιουργικότητά μας και κυρίως θέλουμε να προσφέρουμε περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες στα παιδιά μας, τις νέες γενιές, περισσότερες θέσεις εργασίας, καλύτερες, καλύτερα αμοιβόμενε. Αυτό είναι το InvestEU. Πάνω και πέρα από αριθμούς, αν και βεβαίως έχουν και οι αριθμοί την αξία τους. Ο στόχος του προγράμματος που εκτείνεται από το 2021 έως το 2027 είναι να προσελκυστούν επενδύσεις 650 δισεκατομμυρίων ευρώ, να δημιουργηθούν εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας και να χρηματοδοτηθούν επίσης δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με βάση τη νέως τώρα εφαρμογή του EFCI του επενδυτικού προγράμματος που εκτιμάται ότι μέχρι το 2020 θα φέρει επενδύσεις ύψους 500 δις ευρώ, θα χρηματοδοτήσει 850.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα συμβάλλει στη δημιουργία 1,4 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, δικαιούμαστε με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση να θέσουμε τον πύχη των προσδοκιών ακόμη ψηλότερα. Για παράδειγμα, όσον αφορά το συνολικό ύψος των επενδύσεων. Προσωπικά εκτιμώ ότι με το InvestEU θα προσεγγίσουν το 1-3 ευρώ και πρόκειται να δημιουργηθούν πάνω από 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Άλλωστε, έχουμε πλέον την εμπειρία από την εφαρμογή του EFCI και είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τι χρειάζεται να διατηρήσουμε και τι να βελτιώσουμε ή να αλλάξουμε. Προς την κατεύθυνση αυτή φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας, η οποία είναι προϊόν συστηματικής και επίπονης εργασίας, αλλά και εκτεταμένου διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τους εκπροσώπους δεκάδων φορέων κοινωνικών, επιχειρηματικών και φυσικά αυτοδιοικητικών από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη γνωμοδότησή μας αναδεικνύουμε ως πρώτη της σημασίας να συμπεριλαμβάνεται στους στόχους του προγράμματος η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ευρώπης η ευρωπαϊκή επιτροπή εκτιμά ότι το 2021 το ακαθάριστο εθνικό προϊόν στις περισσότερες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης θα έχει ανέλθει στα προκρίσης επίπεδα. γι' αυτό αποδίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στο να είναι το γεωγραφικά ισορροπημένο και να στοχεύει κατά προτεραιότητα στις περιφέρειες που πάσχουν από ουσιαστικέ και χρόνιες ελλείψεις επενδύσεων προτείνουμε με έμφαση το πρόγραμμα να εφαρμοστεί μέσω της στενής συνεργασίας με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές οι οποίες όπως φυσικά και η επιτροπή περιφερειών πρέπει να έχουν λόγο ώστε να φτάσουμε σε καλύτερα αποτελέσματα και κυρίως στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο να εφαρμοστεί το πρόγραμμα με ταχύτητα, χωρίς αχρίαστες γραφειοκρατικές διαδικασίες και βεβαίως αφού βεβαίως διασφαλιστεί ότι η ταχύτητα δεν θα επηρεάζει την ποιότητα των αποφάσεων αυτών, αλλά και την ποιότητα των έργων. Τονίζουμε ότι το InvestEU είναι ένα πολυεργαλείο για τη δημιουργία νέων, καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι η ρεχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, την προσέλκυση επενδύσεων και μάλιστα σε νευραλικές υποδομές αλλά σε υποδομές του κοινωνικού τομέα. Την προστασία του περιβάλλοντος, την αποφασιστικότερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την υποστήριξη υπηρεσιών που εντάσσονται στο κοινωνικό κράτος, το σημαντικότερο επίτευγμα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ενθάρρυνση της καινοτομίας, την επιτάχυνση της ψηφιακής σύγκλησης, την υποστήριξη της έρευνας. Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη ήταν πάντοτε στην πρωτοπορία. Τα τελευταία χρόνια δέχεται έντονο ανταγωνισμό από άλλες υπήρους και άλλες χώρες. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πλανήτη και να μας περιμένει να ανεβούμε. Χρειάζεται να ανακτήσουμε ξανά την πρωτοβουλία των κινήσεων, να ξαναγίνουμε πρωτοπόροι στην οικονομία, την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, ενώ παράλληλα διατηρούμε την πρωτοπορία σε πολιτικές με κυρίαρχη αυτή την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της κοινωνικής προστασίας. Εξασφαλίζουμε ένα ισχυρό δίκτυο κοινωνικής προστασίας για κάθε Ευρωπαία, για κάθε Ευρωπαίο. Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη του μέλλοντος χρειάζεται innovators, disruptors και above all doers. Be the change, let's be the change. Ας είμαστε εμείς η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν παρεμβάσεις μέσα στα πλαίσια της γενικής συζήτησης. Φαίνεται πως όχι. Φτάνουμε λοιπόν στις τροπολογίες. Προτείνω να, τις, να ψηφίσουμε μία με έξι από κοινού υπέρ. Κατά εγκρίνονται. Προτείνω ψηφοφορία unblock για τις 7 και 9 υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Le vote est clos. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία. Προτείνω να ψηφίσουμε unblock τις 8, 10 και 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Προτείνω ψηφοφορία unblock για τις 12 και 13. Υπέρ κατά εγκρίνονται 14 υπέρ κατά εγκρίνεται 15 υπέρ κατά απορρίπτεται 16 υπέρ κατά εγκρίνεται unblock 17-18 υπέρ κατά εγκρίνονται 19 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 20 υπέρ κατά απορρίπτεται τώρα τελική ψηφοφορία υπέρ της γνωμοδότησης παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται το έγγραφο ομόφωνα να συγχαρούμε τον συντάκτη και την ομάδα του. Τώρα, το πρόγραμμα στήριξη μεταρρυθμίσεων και λειτουργία ε, σταθεροποίησης επενδύσεων. Όλγα Σρίεν. Η έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το πρόγραμμα αυτό στήριξης μεταρρυθμίσεων και σταθεροποίησης επενδύσεων έχει 25 εκατομμύρια ευρώ συνολικά και ελπίζουμε να υποστηρίξει τις κατά προτεραιότητα μεταρρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρία στοιχεία θα πρέπει να τονιστούν. Καταρχήν ε, ότι θα πρέπει να υπάρχει μία υποστήριξη μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με 22 δις ευρώ που να διαθέτουν όλα τα κράτη-μέλη. Ένα μέσο τεχνικής υποστήριξης για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τις μεταρρυθμίσεις και τη διοικητική τους ικανότητα. Και αυτό βασίζεται στην πείρα της ομάδας υποστήριξης η οποία την τελευταία φορά ενέκρινε 440 ε, προγράμματα τα τελευταία χρόνια. Ένα μέσο που να διαθέτουν όλα τα κράτη-μέλη με προϋπολογισμό 0,94 ε, δις ευρώ και επίσης προϋπολογισμό 16 ε, δις ευρώ μέσα στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης για τα κράτη τα οποία έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα εισήγησης της Ευρωζώνης. Πρόκειται για ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ολικής στήριξης. Οι προτάσεις που εδώ αναγράφονται λαμβάνουν υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και με βάση αυτή την αρχή το πεδίο εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων αφορά τους στρατηγικούς ε, τομείς για την εφαρμογή των ε, ε, διατάξεων της συνθήκης και των προσταγών της συνθήκης. Δεν δεχόμαστε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που δεν είναι εξειδικευμένες και που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης και που επίσης δεν συνεισφέρουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν διευρύνουν τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δείκτες που εγκρίνονται σε σχέση με την πολιτική συνοχής για την περίοδο 21-27. Σας υπενθυμίζω ότι πρόκειται για το, ΑΕΠ, για το κατακεφαλή ΑΕΠ, τη συνοχή, την ανεργία των νέων, την εκπαίδευση, τις κλιματικές αλλαγές, την υποδοχή και την ενσωμάτωση των ε, μεταναστών, όλα αυτά θα πρέπει να έχουν σωστή κλίδα κατανομής. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει μία συνοχή και επίσης να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι οι ανάγκες μεταρρύθμισης για ορισμένα κράτη αφορούν 7 απτά μέτρα για να μπουν στην Ευρωζώνη κάτι το οποίο είναι επιτακτικής, θέμα επιτακτικής ανάγκης σε σχέση με την Ευρωζώνη. Ως προς το θέμα μεταφορών, το πρόγραμμα στήριξης μεταρρυθμίσεων δεν είναι ένα επενδυτικό ε, πρόγραμμα με βάση το πρόγραμμα και το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Άρα θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε έναν υψηλό κίνδυνο ε, απόρριψης εάν διατηρηθεί η ικανότητα μεταφοράς. Γι' αυτό δεν θα θέλαμε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα μεταφοράς. Θέλουμε μια αιτιώδη συνάφεια με το ευρωπαϊκό εξάμεινο έτσι ώστε να υποστηριχτούν οι αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις. Και επίσης θα θέλαμε οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να ενισχυθούν μέσα στα πλαίσια της διοικητικής τους επάρκειας, γιατί αυτό ήταν ένας αδύναμος κρίκος. Μια προσέγγιση λοιπόν η οποία συνάδει με τις ανάγκες της ε, Επιτροπής των Περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή ανάπτυξη. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω την εξαιρετική εργασία στα πλαίσια του προγράμματος μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την κυρία Αμπάλ και την κυρία Ναρτίγαλ. Και οι δύο έλαβαν υπόψη τα δικά μας αιτήματα και θα προωθήσουν τα προγράμματα αυτά και τα κείμενα υπό αυτή την έννοια. Μέσα στα πλαίσια των input ήρθαμε σε επαφή και με την ΕΟΚΕ, η οποία μας άκουσε πολύ προσεκτικά σε σχέση με την ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Η εργασία αυτή είναι τεχνική υφής, αλλά ουσιώδους σημασίας και είδαμε ότι υπάρχει θέληση συνοχής και διαφάνειας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και προς τη Γραμματεία και προς τον εμπειρογνώμονά μου, χωρίς την συνδρομή του οποίου δεν θα ήταν δυνατή αυτή η εργασία. Ποιος θα ήθελε το λόγο. Δεν βλέπω κανείς να ζητά το λόγο. Φτάνουμε λοιπόν στις τροπολογίες. Προτείνω ψηφοφορία unblock για την 1 και 3 υπέρ κατά εγκρίνονται. Δύο υπέρ κατά απορρίπτεται. Ψηφοφορία unblock για τις 4 και 7 υπέρ παρακαλώ κατά εγκρίνονται. 5. 5. Άρα εκπίπτει 6 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8. Άρα καταπίπτει 9 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. κατά, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία επί της γνωμοδότησης, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Με μεγάλη πλειοψηφία να συγχαρούμε την εισηγήτρια και την ομάδα της. Περνάμε τώρα στην γνωμοδότηση όσον αφορά το πακέτο για την ε, δέσμη μέτρο, μάλλον για την ε, διεύρυνση. Ο Φράνκο Ιάκοπ έχει το λόγο. Monsieur le rapporteur, vous avez la... Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εκπόνηση της γνωμοδότησης αυτής την όλη υποστήριξη που είχα από τη Γραμματεία και από τον εμπειρογνώμονά μου. Καθώς επίσης να ευχαριστήσω και όλες τις ε, αρχές και τις θεσμικές αρχές, να ευχαριστήσω επίσης την Προεδρία την Ευρωπαϊκή της Αυστρίας και της Βουλγαρίας, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και τους πρέσβει από τις υποψήφιες προσένταξη ένταξη χώρες, αλλά και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες, καθώς επίσης και όλους τους οργανισμούς περιφερειακής συνεργασίας, καθώς επίσης και τα τοπικά περιφερειακά δίκτυα, τα οποία υφίστανται για την περιφερειακή συνεργασία στις χώρες αυτής. Το λέω αυτό διότι Κατά την εκπόνηση της γνωμοδότησης αυτής έπρεπε να γίνουν και συνεχείς προσαρμογές καθότι εξελισσόταν και η πολιτική κατάσταση των χωρών αυτών και καθότι εγκρίνονταν στο ενδιάμεσο διάστημα διάφορες αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για παράδειγμα, το Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου είπε ότι η Αλβανία, η πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μπορούν να πάρουν ήδη το 19 μια μερομηνία ένταξης έναρξη διαπραγματεύσεων. Έχουμε την ιστορική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για την ονομασία όπου μπορεί η διαδικασία να μην έχει ακόμα ολοκληρωθεί, αλλά βρίσκεται στα πλαίσια κοινοβουλευτική ανάλυση και εξέταση από την πλευρά τη ΦΥΡΟΜ. Έχουμε επίσης εξελίξεις και σε άλλες χώρες, όπως και στην Τουρκία, όπου βέβαια η κατάσταση δεν έχει ομαλοποιηθεί. Έχουμε και τις εκλογές στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, όπου είχαμε μια θετική εξέλιξη όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό και την ειρήνευση στην χώρα αυτή. Το σχέδιο επίσης γνωμοδότησης συζητήθηκε τον Σεπτέμβριο στην Επιτροπή ΣΥΒΕΞ Έγινε μια πολύ ειλικρινή συζήτηση με διάφορους συναδέλφους. Είχαμε κατά αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να ενσωματώσουμε όλες τις προτινόμενες τροπολογίες. Στη γνωμοδότησή μου αυτή εν γέννη λέω ότι η διεύρυνση θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κράτος δικαίου, δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν προφανώς αναπόσπαστα στοιχεία της όλης αυτής διαδικασίας η δέσμοι μέτρων για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μα βρίσκει σύμφωνους, αλλά λέμε στη γνωμοδότηση αυτή ότι δεν δίδεται αρκετή σημασία και βάρος στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν και διαδραματίσουν τοπικές και περιφερειακές αρχές. Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το λένε και οι συνάδελφοι αυτοί που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας επαφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψηφίων αυτών κρατών. Λέμε ότι το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό τονίστηκε σε όλες τις ε, συναντήσεις που είχαμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να μπορεί να συμβάλλει γενικότερα στη διεύρυνση. Είμαστε πεπισμένοι ότι η διεύρυνση θα πρέπει να είναι μια διεύρυνση κοινοτήτων, μια διεύρυνση των ίδιων των πολιτών. Θα πρέπει να ξεκινά από το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Δεν μπορεί να είναι απλώ ένα εγχείρημα το οποίο θα λαμβάνει η χώρα μόνο σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο. Θα πρέπει πραγματικά να δίνονται πάρα πολλέ δυνατότητε μέσω τη διεύρυνση και στου ίδιου του πολίτε. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο θέλουμε να ενισχύσουμε τα όργανα και τα εργαλεία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψηφίων ή δυνάμει υποψηφίων χωρών. Θέλουμε όμω η συνεργασία αυτή να γίνεται και σε τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να προωθήσουμε προγράμματα όπως το ΣΥΓΜΑ ή τα προγράμματα αδελφοποίηση. Θέλουμε να ξεκινήσει επίσης εκ νέου να χρηματοδοτείται ο μηχανισμός για την αυτοδιοίκηση, το Local Administration Facility και θέλουμε να έχουμε και μία ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να μπορούμε να έχουμε πραγματικές γνώσεις και διοικητικές ικανότητες σε επίπεδο τοπικής, αυτοδιοίκηση. τοπικής αυτοδιοίκησης. Λέμε επίσης στη γνωμοδότηση αυτή ότι προφανώς αναδύονται νέες ευκαιρίες μέσω της διαδικασίας της διεύρυνσης Λέμε επίση ότι είναι πολύ θετική στάση που κρατάει η Σερβία και η Τουρκία όσον αφορά τη διαχείριση τη ροή των μεταναστών. Ήδη έχουν αντιληφθεί πολλέ θετικέ δράσει, αλλά η επιτυχία των δράσεων αυτών έχει να κάνει και με την ικανότητα που έχουν σε διοικητικό επίπεδο οι περιφερειακέ και τοπικέ αρχέ. Λέμε επίση ότι θα πρέπει από κοινού να προστατεύσουμε το την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά όλων των χωρών. Τώρα, όσον αφορά κάποια πιο συγκεκριμένα σημεία, θεωρούμε ότι για τα Δυτικά Βαλκάνια υπάρχουν και δυνατά και αδύναμα σημεία σε εθνικό επίπεδο και λέμε ότι η διαδικασία της διεύρυνσης που θα πρέπει να προωθηθεί αποφασιστικά ήδη από το 2018 και μέσα στο 2019 αποτελεί ουσιαστικά μια ευκαιρία. Είναι κρίμα όμως να βλέπουμε ότι σε ορισμένες χώρες υπάρχει μια κάποια απεσιοδοξία και ένα σκεπτικισμός απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο λέμε στη γνωμοδότηση αυτή, αναφερόμενη κυρίως στην Τουρκία, ότι αυτό που έχει αρχίσει να φαίνεται εδώ και κάποιο καιρό ως μια απομάκρυνση της Τουρκίας από την ευρωπαϊκή προοπτική θα πρέπει να αντίστραφει εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει η Τουρκία να ακολουθήσει την ευρωπαϊκή αυτή πορεία που ξεκίνησε στο παρελθόν. Ξέρουμε ότι η Τουρκία πρόσφατα ενέκρινε αυτό το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, το οποίο επιβαρύνει ιδιαίτερα τις δημοκρατικές διαδικασίες σε τοπικό επίπεδο. πρόεδρος πρέπει να ολοκληρώσει, παρακαλώ πολύ, έχετε ήδη υπερβεί κατά πολύ το χρόνο αγόρευσή σας. Τελευταία παρατήρηση κάνω, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την Σερβία λέμε ότι εδώ έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις, ιδίως όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση στη Βοηδοβίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Ποιος θέλει το λόγο στα πλαίσια της γενικής συζήτησης, λέει ο Πρόεδρος. Ουδής. Λοιπόν, ας περάσουμε τότε ευθύ αμέσω στις τροπολογίες. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 2 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 του συγητή που αντικαθιστά την 3 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 του συγητή που αντικαθιστά την 4 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά απορρίπτεται. Μαζί τις 7 έως 11 ψηφίζουμε υπέρ παρακαλώ, κατά εγκρίνονται. Περνάμε έτσι στην τελική ψηφοφορία για το στόλο της εκδομοδότησης υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές. Η γνωμοδότηση γκρίνεται ομόφωνα Συγχαρητήρια στον εισηγητή και στην ομάδα του. Nous Ας περάσουμε τώρα στην γνωμοδότηση του συναδέλφου Jean-Luc Varnas όσον αφορά τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Monsieur le rapporteur, Κύριε Ισηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, επιτρέψτε μου να έρθω σύντομα ε, στην ανάπτυξη του προβλήματος. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Σε ορισμένες επιχειρήσεις και ιδίω αυτές που δραστηριοποιούνται στον ψηφιακό τομέα αυτές λοιπόν πληρώνουν ελάχιστου φόρους και έτσι προκαλείται ένα αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι ιδίω στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες τελικώς αναλογικά πληρώνουν πολύ μεγαλύτερου φόρους. Πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται όπω είπα στον ψηφιακό τομέα και χρησιμοποιούν ψηφιακά συστήματα, προσφέρουν ψηφιακές υπηρεσίες και φαίνεται πως διάφορες χώρες στην Ευρώπη έχουν αναλάβει τώρα την πρωτοβουλία να καθορίσουν ιδίους φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι όμως διαφέρουν μεταξύ τους. Εξετάσαμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ίσως θα πρέπει να αναλυφθεί άλλη πρωτοβουλία από την οποία να προκύπτει εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών. Διότι ε, προκειμένου δεν ενδιαφέρει να καθορίζουν οι επιμέρους χώρες μέλη δικούς τους φορολογικούς συντελεστές, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι εναρμόνιση. Πρέπει να ληφθούν βέβαια υπόψη ορισμένα πράγματα. Πρέπει να αποφευθεί η διπλή φορολόγηση. Επίσης, το πεδίο εφαρμογή ε, του εν λόγω φόρου πρέπει να προσαρμοστεί στις ε, διάφορες επιχειρήσεις. Αυτά θα τα δούμε. Αλλά επίσης σημαντικό είναι ότι Ορισμένες επιχειρήσεις του ψηφιακού τομέα λειτουργούν ε, με ζημία. Όμως αυτό δεν επηρεάζει πολύ την φορολόγηση εφόσον έχουν ε, άνω της ε, δεκαετίας δραστηριότητες. Το ερώτημα είναι τώρα και εάν μπορεί να γίνει φορολόγηση στον τόπο που προσφέρεται η υπηρεσία. Εκεί δηλαδή όπου ο καταναλωτής καταναλώνει το σχετικό προϊόν ή υπηρεσία προσφέρει η επιχείρηση. επιχειρηση υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα και ένα από τα μέτρα αυτά είναι ναι, το κριτήριο της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας. Και εδώ βεβαίως πρέπει να γίνουν οι σχετικές προσαρμογές. Υπάρχουν διάφορες λύσεις που προτείνονται. Μία ε, βραχυπρόθεσμη λύση και οι περισσότερες επιχειρήσεις με τις οποίες ε, συνομίλησα φαίνεται να δηλώνουν ικανοποιημένες. Υπάρχει και μια μακροπρόθεσμη λύση που φαίνεται πως είναι πιο δύσκολη. Πάντως το καλό νέο είναι ότι ο ΩΣΑ θα εγκύψει το θέμα ε, ήδη από το 2020 ο ΣΑ έχει κάνει μια σχετική προεργασία για την αποφυγή της φοροαποφυγής, για την αποτροπή καλύτερα της φοροαποφυγής και αναφέρομαι στο σύστημα ή μάλλον στο σύστημα αποφυγής των BEPS και βέβαια πρέπει να απολύξει η προσπάθεια αυτή σε μια φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών. Το 2020-2021 θα πρέπει να λάβει η φορολογία αυτή μια τελική μορφή ε, που να συμβαδίζει και με τις συμφωνίες που συνάπτονται στον ΟΟΣΑ. Τίθεται ορισμένα ερωτήματα. Είναι καλή η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών και επίσης για το γεγονός ότι όλα τα κέρδη από δραστηριότητες των επιχειρήσεων θα φορολογούνται εκεί όπου γίνεται η κατανάλωση των ε, σχετικών υπηρεσιών. Βράχει πρόθεσμα, η λύση μπορεί να δοθεί και υπό την παρούσα Προεδρία. Αλλά την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίθηκε η σχετική έκθεση και παρακαλώ να εγκρίνετε και τη σημερινή μας γνωμοδότηση μαζί με τις παρατηρήσεις τις οποίες μόλις σας υπέβαλα ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ φίλε και ιδίω για τον σεβασμό του χρόνου αγορεύσεως σπάνιο και γι' αυτό το τονίζω. Ποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο τώρα στην γενική συζήτηση. Je ne vois pas de demande, alors nous... Ε, δεν βλέπω κανένα να ζητεί. Ερχόμαστε λοιπόν στις τροπολογίες και προτείνω να ψηφιστούν όλες μαζί ή 1, 2 του εισηγητού που αν ψηφιστούν εκπίπτουν η 4, 1 και η 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται οι τροπολογίες. Η τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Όχι, καλύτερα να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. vote. Πέρας της ψήφου. Απερίφθη η τροπολογία. Τροπολογία υπαρθών 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία υπέρ της γνωμοδοτήσεως. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με πάντως πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά και σας ευχαριστούμε για την εργασία σας. Τώρα ακολουθεί γνωμοδότηση για την χρηματοδότηση της αηφόρου ανάπτυξης με εισηγητή τον κύριο Γκούντλακ. Non, non, non, la résolution. trop vite avec la résolution. jamais. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Έχει το λόγο κύριε Σιγητά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξιότιμες κύριε και κύριοι, έχω σήμερα την χαρά να σας παρουσιάσω το σχέδιο δράσης για τη χρηματοδότηση αηφόρου ανάπτυξη. Οι πρωτοβουλίε αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ πλαίσιο προώθησης ε, στόχων αηφόρου ανάπτυξη. κάτι που είναι απολύτω επίγον. Οι ειδικοί διαπιστώνουν ότι αύξηση, η αναμενόμενη αύξηση της θερμοκρασίας θα είναι της τάξης των 3,2 βαθμών, 3,2 βαθμών. Άρα δεν μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του Παρισιού. Ούτως ή άλλως, άλλωστε έχουμε ξεπεράσει ήδη τους 1,5 βαθμούς του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κλίματος είναι τεράστια η δυναμική της αλλαγής του κλίματος και φαίνεται στο, στους πάγους του Βόρειου Πόλου, η οποία από το 1998 έχει μειωθεί κατά 36%. Άρα πρέπει να δοθούν σοβαρά κίνητρα για την χρηματοδότηση αηφόρου αναπτύξεως και οι ροές κεφαλαίου πρέπει να κατευθυνθούν προς βιώσιμες επενδύσεις. Ένας, μία οδός μπορεί να είναι μέσω του χρηματοδοτικού συστήματος και κυρίως για να αποφευθεί η απατηλή επισήμανση των έργων, δηλαδή να παρουσιάζονται ως βιώσιμα ενώ δεν είναι. Σε όλες τις στρατηγικές της Ένωσης πρέπει να περιλαμβάνονται οι στόχοι της βιωσιμότητας. Η γνωμοδότηση που σας υποβάλλουμε υποστηρίζει τις προσπάθειες δημόσιων και ιδιωτικών επενδυτών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των αλλαγών του κλίματος και της βιωσιμότητας και για να καλυφθεί το τεράστιο κενό επενδύσεων στο κλίμα και για να υπάρξει εμπιστοσύνη και περισσότερη διαφάνεια διότι ως τώρα δεν υπάρχει σαφήνεια εάν οι παράγοντες, κοινωνικοί παράγοντες και οι παράγοντες governance περιλαμβάνονται όντως τις αποφάσεις για τις επενδύσεις. Το άλλο θέμα είναι η αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών κινδύνων που προέρχονται από τις ε, επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος που ήδη ε, απειλεί με σημαντικές οικονομικές ζημίες. Ένα ρόλο παίζει και η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος με την έννοια της ε, Ένωσης Κεφαλαίων. Το σχέδιο περιλαμβάνει ως βασικό βήμα τη δημιουργία συστήματος ταξινόμησης για βιώσιμες επενδύσεις. Την άνοιξη του 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει κατάλογο κριτηρίων για βιώσιμες επενδύσεις. Θα καταλήξουμε έτσι να χρησιμοποιούμε μια κοινή γλώσσα σχετικά με το ποιε επενδύσει μπορούν να χαρακτηριστούν βιώσιμε. Και αυτό θα αποτελέσει τη βάση για άλλε δραστηριότητε όπω θέσπιση προτύπων κλπ με την χρηματοδότηση τότε των επενδύσεων αυτών θα είναι δυνατόν να αρχίσουμε για να ενισχυθούν οι σχετικές δραστηριότητες. Είναι σαφές ότι δεν αρκούν βεβαίω αυτά. Η βιωσιμότητα για μένα είναι κάτι παραπάνω από το πράσινο χρώμα. Το έτσι βλέπει τα πράγματα και η τράπεζα Κάριτας. Δεν η βιωσιμότητα είναι αίτημα παγκόσμια ισχύω και στηρίζεται και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με τους ε, βιώσιμους στόχους ανάπτυξης που έχουν θεσπίσει και προβάλλουν για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της σημερινής γενεάς χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι μελλοντικέ γενναίες. Γνωρίζουμε τις ε, προσπάθειες του επιχειρηματικού και ασφαλιστικού κόσμου να ε, στραφεί προς πιο βιώσιμες επενδύσεις και αυτές ενισχύονται από την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ζήτηση για πράσινες επενδύσεις αυξάνεται παγκόσμια, αλλά δεν υπάρχουν ακόμα τα ξεκάθαρα κριτήρια για το τι σημαίνει πράσινη δανειοδότηση. Κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξουν τα κριτήρια αυτά. Και πράγματι για να υπάρξουν και ανθρώπινες αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και για την παραγωγή και για την διάθεση στην εμπορία. Είναι σημαντικές οι ευθύνε που πρέπει να αναλυθούν ώστε τα χρησιμοποιούμενα benchmark να σέβονται, για παράδειγμα, και τον στόχο των δύο βαθμών Κελσίου. Πρέπει να είναι σαφές για τους επενδυτές τι υποστηρίζουν με τα χρήματα που διαθέτουν για επενδύσει. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Αρχίζει η γενική συζήτηση. Έχω ήδη έναν συνάδελφο που ζητεί το λόγο, ο κύριος Μαρτίνες Αρεγκουή. Κύριε Πρόεδρε, κύριε εισηγητά, θα ήθελα να λάβετε υπόψη την τροπολογία συμβασμού σε σχέση με την αηφόρο ανάπτυξη πέρα από αυτό τον πολιτικό συμβιβασμό πρόκειται για ένα νομικό μέσο έτσι ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτές τις επενδύσεις για τη βιωσιμότητα. Νομίζω ότι ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μία αρχή, αλλά αναφέρεται αποκλειστικά στις οικολογικές πράσινες πτυχές και τις πτυχές του περιβάλλοντος και έχει ξεχάσει όλη την κοινωνική πτυχή, τη... καθώς και την απασχολησιμότητα για να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα φυσικά. Ε, εμείς φέρουμε μεγάλη ευθύνη ως περιφερειακές αρχές για τις επενδύσεις στη βιομηχανία, στα ύδατα, στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, αλλά υπάρχουν και πολλές δαπάνες στο τομέα της απασχόλησης, ε, της κοινωνικής ανάπτυξης και της υγείας. Θα θέλαμε πραγματικά να προωθηθούν αυτοί οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, έχει πολύ μεγάλη σημασία η ύπαρξη δικτών που θα πρέπει να είναι κοινή για όλες τις χώρες έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να μετρήσουμε αυτές τις επενδύσεις που στοχεύουν στη βιωσιμότητα έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις δεσμεύσεις έμπρακτα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κριστό Φρουγιόν έχει το λόγο. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή για την ποιότητα της εργασίας του. Θα πρέπει να βρούμε τη λύση για να συνδυάσουμε το θέμα της αγοραστικής δύναμης και της προστασίας του πλανήτη, καθώς και τις βιώσιμες επενδύσεις, τις επενδύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη προς τα πάνω και για να ε, ξεφύγουμε από το δημοσιονομικό αδιέξοδο που κατασπαταλά το δημόσιο χρήμα φτάνοντας σε μια ολική νέκρωση με βάση τη χρήση κυρίως του άνθρακα. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από την οικονομία του άνθρακα για να μην καταστραφεί ο πλανήτης, και να βρούμε και μια λύση για τους συμπολίτε που με δυσκολία τα βγάζουν πέρα μέχρι το τέλος του μήνα. Δεν ζητά κανένας άλλο το λόγο, γι' αυτό μπορούμε τώρα να περάσουμε στην ψηφοφορία των τροπολογιών. Προτείνω να ψηφίσουμε on block τις 1 και 3 υπέρ. Κατά εγκρίνονται 2 υπέρ κατά, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε on block τις 5 και 6 υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 7 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία επί της γνωμοδότησης υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται ομόφωνα και να συγχαρούμε τον εισηγητή και την ομάδα του. Τώρα, περνάμε στην γνωμοδότηση για τα πρότυπα τοπικής ενεργειακής ιδιοκτησίας και το ρόλο των τοπικών κοινοτήτων στην ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη. Πρόκειται για γνωμοδότηση πρωτοβουλίας που θα μας παρουσιάσει η εισηγήτρια Μαριάννα Γκάζου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να σας απευθύνω το λόγο σήμερα όπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορέσαμε να γιορτάσουμε την ημέρα της Μεγάλης Ένωσης της Ρουμανίας. Εμείς, οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών που είμαστε υπεύθυνοι για τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές, θα πρέπει να σας παρουσιάσουμε μία γνωμοδότηση που αφορά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στις περιφερειακές αρχές και την ποιότητα ζωής των πολιτών που εκπροσωπούμε, καθώς και την ανάπτυξη της εθνικής ε, οικονομίας μέσα στα πλαίσια τιμών ενέργειας που να είναι προσιτές. Η τοπική ενεργειακή αγορά δίνει τα μέσα διαχείρισης της ενέργειας σε επίπεδο κοινότητας με την σωστή διανομή και κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να γίνει μέσω ενεργειακών πόρων που διαθέτουν οι ίδιες οι τοπικές αρχές. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να συμπληρώσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές μέσω εξειδικευμένων στόχων και με την συνεισφορά των τοπικών αρχών σε σχέση με τη χρήση της ενέργειας, πολλές ε, πόλεις συμμετέχουν σε αυτή τη διάσκεψη δημάρχων όπου γίνεται λόγος για την βιώσιμη χρήση ενέργειας. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτός ο στόχος αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές χρήσης το, της ενέργειας και την πολιτική όθηση έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να προωθήσουν τον ε, ρόλο των ε, ενεργειακών τοπικών αρχών. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, διότι κύρωσε αυτή τη φάση της ενεργειακής απόδοσης μέσα στα πλαίσια της εργασίας της. Ευχαριστώ την Επιτροπή Περιβάλλοντος και τους συντονιστές. Αυτή την περίοδο διαπιστώσαμε το εξής. Οι τοπικές αρχές χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους χρήσης της ενέργειας μέσα στα πλαίσια εταιρικών σχέσεων ή μέσω εταιριών περιορισμένης ευθύνης καθώς και οργανισμών που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έτσι, οι τοπικές αρχές μπορεί, μπορούν να μετέρχονται όλων αυτών των μέσων και συνεπώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε σωστά τις ενεργειακές πηγές σε τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και δημοσιονομικά ευεργετήματα, περιορίζοντας την ενεργειακή παινία. Γι' αυτό οι τοπικές αρχές για την ενέργεια ασχολούνται με την αρχή εκδημοκρατισμού, θα μπορούσα να πω, της χρήσης των ενεργειακών πηγών. Έτσι, οι επιχειρηματίες και οι καταναλωτές μπορούν να αναλάβουν ένα πιο σημαντικό ρόλο για, για τη διαχείριση της ενέργειας και αυτό έχει σχέση με τους κοινωνικούς στόχους καθώς και τους περιβαλλοντικούς. Πρέπει να έχουμε ένα καθαρό περιβάλλον, πρωτίστως για τα παιδιά μας που είναι και το μέλλον μας. Επίσης, θα πρέπει να συμμετέχουν ένα και περισσότερο οι πολίτες στη διαχείριση της χρήσης των ενεργειακών πηγών για να ευεργετούνται περισσότερο και να την χάνουν της ε, υποστήριξης της κοινή γνώμης. Ορισμένες τοπικές αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν αυτές τις βέλτιστες ε, πρακτικές και στην Αυστρία η Επιτροπή Περιβάλλοντος έδειξε ποια μπορεί να είναι τα απτά αποτελέσματα ενός τέτοιου προγράμματος έτσι ώστε οι τοπικές αρχές να εξοικονομήσουν χρήματα τα οποία μπορούν να επανεπενδύσουν σε άλλα προγράμματα, διαρθρωτικά προγράμματα καθώς και ερευνητικά. Εμείς προτείνουμε μία σειρά συστάσεων. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας στον τομέα της ενέργειας σε τοπικό επίπεδο και αυτό αφορά ιδιαίτερα τις ανανεώσιμες καθώς και την ενεργειακή μετάβαση με υποστηρικτικούς μηχανισμούς. Παράλληλα θα ήθελα να σας πω ότι προτάθηκαν οκτώ τροπολογίες με την πλειοψηφία συμφωνώ. Αντιτίθεμαι σε δύο. Πρόκειται για την υπαριθμόν 6 που είναι πολύ περιοριστική και δεν αναφέρεται στον μηχανισμό χρηματοδοτικής υποστήριξης. Επίσης, αντιτίθεμε και στην τροπολογία 8, που είναι πολύ περιοριστική ως προς την προστασία των δικτύων. Θα πρέπει λοιπόν να μειώσουμε τον ε, τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα πολλών δικτύων που υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ποιος θα ήθελε να λάβει το λόγο στη συζήτηση. Δεν βλέπω να ζητά κανείς το λόγο. Λοιπόν, περνάμε στις τροπολογίες. Προτείνω ψηφοφορία on block για τις 1 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 6 υπέρ κατά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Le vote est clôturé et l'amendement. Πέρας και απορρίπτεται η τροπολογία. Τροπολογία 7 υπέρ κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας και απορρίπτεται η τροπολογία. Ψηφίζουμε την γνωμοδότηση υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με μία αποχή να συγχαρούμε την εισηγήτρια και την ομάδα της. Και σας ευχαριστώ πολύ για την συνολική εργασία. Nous en venons... Περνάμε τώρα στο σημείο 22 της ημερήσιας διάταξης γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσει για την επανεχρησιμοποίηση των υδάτων. Καλώ τον εισηγητή μας, τον κύριο Όλτριχ Βλάσακ, να έρθει εδώ στο Προεδρείο. Κύριε εισηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, πιο συγκεκριμένα για αυτό το οποίο αποκαλούμε νερό από ανάκτηση, ύδατα που ανακτώνται. Το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά λόγω της διψιδρίας, της έλλειψης νερού στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το νερό από ανάκτηση, κυρίως στις γεωργικές καλλιέργειες. Η υφιστάμενη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα αυτό ισχύει και εφαρμόζεται σε έξι μόνο κράτη-μέλη. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να καλύψουμε περαιτέρω το ζήτημα αυτό, προκειμένου να μπορούν και άλλα κρατημέλη να χρησιμοποιούν ανακτώμενο νερό για την άρδευση των καλλιεργειών τους. Το νερό αυτό είναι μόνιμα διαθέσιμο σε αντίθεση με τα υπόγεια ύδατα ή τα επιφανειακά ύδατα, τα οποία εξαφανίζονται όπως ξέρετε σε περίοδους ξηρασίας. Ένας άλλος λόγος χρησιμοποίησης των ανακτώμενων υδάτων είναι ότι ε, κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε κατ' ουσίαν επαναχρησιμοποίηση διαθέσιμου νερού και επομένως δεν θα χρειαστεί κανείς να καταβάλει περισσότερα από σένας γεωργός για παράδειγμα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε μεγαλύτερες ποσότητες ε, νερού. Εξετάζοντας λίγο το όρο σκεπτικό που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή τη, αναφέρεται εδώ πέρα μια ανησυχία που έχει να κάνει με την ασφάλεια των τροφίμων. Και αναφέρει επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ε, επεξεργασμένων λιμάτων για την ε, άρδευση όχι μόνο των καλλιεργειών, αλλά και για την άρδευση αστικών πάρκων, κήπων κτλ. Προσπαθούμε εμείς να καλύψουμε μέσω της γνωμοδότησης αυτής όχι μόνο τους φορείς εκμετάλλευσης των μονάδων ανάκτησης, αλλά και τους χρήστες των υδάτων αυτών. Δύο τροπολογίες έχω λάβει, αγαπητοί συνάδελφοι, για την γνωμοδότηση αυτή. Τη συζητήσαμε τις τροπολογίες αυτές με τους συντάκτες τους και προτείναμε και προφορικές τροπολογίες, ο προτείνω να εγκρίνουμε. Όλες οι υπόλοιπε παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη γνωμοδότηση αυτή έχουν ήδη συμπεριληφθεί στη γνωμοδότηση. Ολοκληρώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονές μου και όλους όσοι συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση και την εκπόνηση αυτής γνωμοδότησης. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ και υποβάλλω μια γνωμοδότηση που πραγματικά ενσωματώνει όλες τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινάει η γενική συζήτηση. Κίρστιν Βίλ, η πρώτη συνάδελφος που θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στο πλαίσιο της κατάρτισης των τροπολογιών. Όσον αφορά τους τελικούς χρήστες των ανακτώμενων αυτών υδάτων, λέγεται εδώ πέρα ότι θα πρέπει να δοθεί άδεια από τις τοπικές αρχές. Με αυτό ισχύει ήδη στη Δανία και θεωρούμε ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί καλά, θετικά, γιατί ουσιαστικά καλούμεθα εδώ πέρα να δούμε πώς αποθηκεύει το ανακτώμενο είδωρο ο τελικός χρήστης και πώς το χρησιμοποιεί. Είναι σημαντικό να υπάρχει δηλαδή μια τοπική εποπτική αρχή όσον αφορά την χρήση των υδάτων αυτών. Δεν αρκεί απλώς να στέλνει κανείς μια ειδοποίηση προς την τοπική αρχή λέγοντας ότι έχει την πρόθεση να επαναχρησιμοποιήσει νερό από ανάκτηση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ λοιπόν για τη συμβαστική τροπολογία επί της οποίας συμφωνήσαμε για την απόκειται πλέον στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν ποιο θα είναι το σύστημα κοινοποίηση και αδειοδότησης όσον αφορά την επανεχρησιμοποίηση των υδάτων. Συμφωνούμε με την τελική μορφή λοιπόν που πήρε αυτή η τροπολογία και θεωρούμε ότι στα πλαίσια της ασφάλειας και της προστασίας των καταναλωτών είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την τροπολογία. Μην ξεχνάμε ότι εμείς στην Δανία είχαμε ακόμα και θανάτους από ανθρώπους που κατανάλωσαν λαχανικά τα οποία είχαν ε, ποτιστεί με μολυσμένο νερό. Πρόεδρος, θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι, επομένως περνάμε στην ψηφοφορία των τροπολογιών. Τροπολογία υπαριθμών 1, όπου εδώ έχουμε και μια συμβιβαστική προφορική τροπολογία. Δίνω το λόγο πάλι λοιπόν για την τροπολογία αυτή στον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να σχολιάσω περαιτέρω την τροπολογία αυτή. Η προλαλήσασα εξήγησε πάρα πολύ καλά το περιεχόμενο αυτή τη τροπολογία. Καταλήξαμε συμφωνία και εναπόκειτο, όπω ακούσαμε, στο κάθε κράτο μέλο να επιλέξουν μεταξύ άδεια επίσημη ή απλή κοινοποίηση. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία υπεριθμών 1 με τη συμβαστική προφορική τροπολογία υπέρ παρακαλώ κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία. Περνάμε στην τροπολογία 2, όπου και εδώ έχουμε μια συμβιβαστική προφορική τροπολογία. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναφερόμαστε στο ίδιο ζήτημα. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία παρελθόν 3 υπέρ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Παρακαλώ για την τροπολογία 3, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 4, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία υπέρ της γνωμοδότησης παρακαλώ. Κατά αποχές. Η γνωμοδότηση εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή και την ομάδα του. Περνάμε τώρα στην γνωμοδότηση του κυρίου Άντρες Γιάγκλα όσον αφορά το διαστημικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα.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 austatud komitee president. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Το διαστημικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό για τις περιφέρειες της πόλης Ευρωπαϊκής Ένωσης, για κάθε Ευρωπαίο πολίτη εν τέλει. Το διαστημικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε όλα τα επιτεύγματα του νέου τεχνολογικού ψηφιακού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους. Είδαμε ότι υπήρχε έντονη εμπλοκή από τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών από πάρα πολλούς παράγοντες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ένα πρόγραμμα πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Μπορεί να μην το συνειδητοποιούμε σήμερα, αλλά οι εξελίξεις στον διαστημικό τομέα ουσιαστικά επηρεάζουν τη ζωή του καθενό. Χάρη στι τεχνολογικέ αυτέ εξελίξει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλε αυτέ τι νέε ευφυεί συσκευέ, τα κινητά τηλέφωνα, καθώ επίση και όλα τα πλεονεκτήματα του νέου ψηφιακού κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη χρησιμοποιεί την διαστημική τεχνολογία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χρησιμοποιούμε τα προγράμματα Κοπέρνικου, Γαλιλαίου και Έγνο. Προγράμματα τα οποία σημείωσαν σημαντικέ επιτυχίε και χάρη στι πρωτοβουλίε αυτέ καταφέραμε να συλλέξουμε πολύ σημαντικά δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τώρα πιο αποτελεσματικά και αποτετικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργήσουμε νέε καινοτόμε υπηρεσίε. Η διαστημική λοιπόν τεχνολογία είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι τεχνολογίες που ε, καθιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πιο αποτελεσματική για συγκεκριμένες ειδικευμένε υπηρεσίες. Δεν έχουμε να κάνουμε λοιπόν μόνο με το διάστημα αυτό καθεαυτό. Ο ιδιωτικό λοιπόν τομέα θα πρέπει να συνεργαστεί με το δημόσιο τομέα όσον αφορά τον τομέα τη διαστημική τεχνολογία και παράλληλα όλα τα αυτά τα νέα δεδομένα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά για το διαδίκτυο των πραγμάτων, για τη γεωργία και για άλλους τομείς. Δυστυχώς είναι περιορισμένη ακόμα η πρόσβαση που έχουμε στα δεδομένα αυτά. Ήδη από το 2016 είχαμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το διάστημα, είχα υποβάλει μάλιστα και μια γνωμοδότηση για την τότε στρατηγική. Τώρα αναφερόμαστε πλέον σε μια πρόταση κανονισμού η οποία ανταποκρίνεται στους νέους στόχους Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το διαστημικό πρόγραμμα και προβλέπονται νέοι στόχοι ενίσχυσης του υφιστάμενου προγράμματος για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων και για τη χρηματοδότηση με 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα νέα αυτά προγράμματα είναι το GovSatCom, το πρόγραμμα για την επιτήρηση και την παρακολούθηση του διαστήματος, καθώς επίσης και προγράμματα εκείνα τα οποία προωθούν περισσότερο την ενημέρωση όσον αφορά το διαστημικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το GovSat.com είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις περιφέρειες. Έχουμε το GNSS, το πρόγραμμα Galileo. Νομίζω όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα να καταφέρουμε να χρησιμοποιούμε περισσότερο το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε το πρόγραμμα Έγνος, ας μην το ξεχνάμε και αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη να εξακολουθήσει να μπορεί να βρίσκει δικές της λύσεις βάσει των νέων αυτών τεχνολογιών. Το πρόγραμμα Galileo δημιουργεί ένα νέο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε επίσης ότι στα πλαίσια της πρότασης αυτής θα δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα. Ήδη όμως έχουμε έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και πολλοί φοβούνται ότι αυτή τη στιγμή ενδεχομένω να υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα είπε ω προ αυτό ότι δεν θα υπάρξουν επικαλύψει και ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί αυτό ο νέο οργανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το διαστημικό πρόγραμμα, γιατί θα επιφέρει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και εμεί αυτό λέμε βέβαια. Όντω θα πρέπει να αποφεληθούμε καλύτερα από τι διαστημικέ τεχνολογίε για να βοηθήσουμε και τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ που μπορούν να αποφεληθούν από τα νέα δεδομένα, καθώ επίση και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Απλώ δεν είναι ξεκάθαρο πώ ακριβώ θα αποφεληθούμε, πώ θα αξιοποιήσουμε τι νέε αυτέ τεχνολογίε. Είναι σημαντικό επίσης η τοπικές και περιφερειακές αρχές να συμμετάσχουν στα λεγόμενα space hubs, τους κόμβους δηλαδή διαστημικής τεχνολογίας που θα δημιουργηθούν, προκειμένου να υποφεληθούν από την νέα αυτή γνώση σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η γεωργία. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε καλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα και τις διαστημικές τεχνολογίες και να δούμε πώς θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε τη νέα αυτή γνώση σε επιχειρηματικό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πρωταρχικό ρόλο στις νέες αυτές διαστημικές τεχνολογίες και είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να συντονίσουμε περισσότερο την διαστημική πολιτική με την πολιτική που ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλου τομεί όπω η ενέργεια, η πολιτική μετριασμού τη κλιματική αλλαγή κ.ο.κ. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα απαραίτητα χρηματοπιστωτικά μέσα για να ενισχύσουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει προκειμένου και αυτές με τη σειρά τους να μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που προκύπτουν από τη διαστημική έρευνα. Το Σεπτέμβριο του 2018 Όταν είχαμε την ε, εκτόξευση ενός νέου πυράβλου που είχε ως ε, προορισμό ένα νέο ε, δορυφορικό σταθμό, αυτό πρόκειται ουσιαστικά για ένα πείραμα το οποίο έκανε η Εστονία, μπόρεσα εκ του σύνεγγυς να παρακολουθήσω την διαδικασία αυτή και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι η δική μου η χώρα, η Αστονία, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη διαστημική έρευνα. Χαίρομαι πάρα πολύ πως μια μικρή πόλη, στην αυτή η οποία εκπροσωπώ, με αρκετού νέους επιστήμονες, κατάφερε και αυτή να εργαστεί και να συμμετάσχει σε μια σε ένα τέτοιο διαστημικό πείραμα και καταφέρνουμε και εμείς να επιφέρουμε τελικά το δικό μας το λιθαράκι, να συμβάλλουμε με το δικό μας το λιθαράκι στην διαστημική αυτή έρευνα που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόεδρε. Ποιος ζητεί τον λόγο. ποιο ζητεί τον λόγο. Εσείς κύριε Βερντόκ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή βεβαίω για την θαυμάσια αυτή γνωμοδότηση την οποία έχει υποβάλει και όπου τονίζει τη σημασία του προγράμματος διαστημικών ερευνών για τις ε, τοπικές κοινότητες και περιφερειακές κοινότητες, κάτι που μας φαίνεται να είναι πάρα πολύ μακριά το διάστημα. Όμως, με την ε, εισήγησή σας καθιστάτε σαφές ποια είναι η σημασία του διαστήματος και για τις ε, πόλεις και περιφέρειες της Ευρώπης. Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Αλλο κανείς δεν βλέπω, λέει ο πρόεδρος. Α, με συγχωρείτε παρακαλώ κύριος Δεκόστερ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ με τη σειρά μου τον εισηγητή για την ποιότητα της εκθέσεως του. Ανέφερε και τον ρόλο που θα πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει πραγματική πρωτοπόρος. Σήμερα για το θέμα του διαστήματο τίθενται τα ίδια ερωτήματα που έθεσαν οι ιδρυτέ πατέρες της Ευρώπη για τον Άνθρακα και το Χάλιβα. Δηλαδή, κοινή προσπάθεια και μια ενιαία κοινή αγορά. Ήδη από το 2009, δηλαδή κοντεύουμε 10 χρόνια πια, έχουμε αρμοδιότητα που ε, δίνει η Συνθήκη της Αβώνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί άραγε για να υπάρξει η διακυβερνητική διάσταση που ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του 80 για θέματα διαστήματος, αλλά και να υπάρξει μια πραγματική φιλοδοξία στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως εδώ και μια δεκαετία δεν έχουμε προχωρήσει. Δεν έχει προχωρήσει ο τρόπος κοινή ας πούμε προσπάθειας, ενώ έχουμε τα αναγκαία μέσα. Σήμερα οι μηχανισμοί που οργανώνουν την διαστημική πολιτική στο ευρωπαϊκό επίπεδο στην πραγματικότητα τροχοπεδούν και μας ε, ξεπερνά ο ιδιωτικός τομέας άλλων υπήρων ενώ γνωρίζουμε ότι Έχουμε εδώ ένα μηχανισμό κυριαρχίας και ένα μηχανισμό ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Επανέρχομαι σε αυτά που λέει ο για να τονίσω και εγώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε πράγματι τα επόμενα χρόνια και να φροντίσουμε να υπάρξει προσέγγιση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να ανοίξουν νέοι δρόμοι και νέοι τρόποι να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής δύναμης στο διάστημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Μάρκ Ράινμαϊστερ. Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και εδώ δημοσίως στην Ολομέλεια δηλαδή, το έχω πράξει ήδη στην ειδική μας επιτροπή, η γνωμοδότησή του είναι εξαιρετική. Το τονίζω και εδώ, διότι το ζήτημα των διαστημικών προγραμμάτων του μέλλοντος έχει ιδιαίτερη σημασία και θα πρέπει να τα πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Γιατί κατά τη γνώμη μου, στον τομέα αυτό, το είπαν και άλλοι πριν, δεν προχωρούμε με επαρκή ταχύτητα. Πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο και να οργανώσουμε καλύτερα το μέλλον. Κάτι ακόμα είναι σημαντικό, όπως το είπε άλλωστε ο κύριος Γιάντλα, το ζήτημα δηλαδή του νέου Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού που πρέπει να αποφύγουμε επικάλυψη με τον υφιστάμενο οργανισμό ESA, European Space Agency. Η δομή της ESA δεν πρέπει να δει να χάνει αρμοδιότητες. Ο Άντρες Ιάδλα τα τόνισε στην έκθεσή του τα πράγματα αυτά και γι' αυτό τον λόγο τον ευχαριστώ και πάλι, διότι περιέλαβε και τις προτάσεις μας αυτές. Και χαίρομαι που θα μπορέσουμε σήμερα να υπερψηφίσουμε το κείμενό του. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Άλλος κανείς, όχι, δεν ζητεί άλλο τον λόγο. Άρα, προχωρούμε στις τροπολογίες. μόνο ένα υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. δύο υπέρ κατά εγκρίνεται Είδου λοιπόν ψηφίστηκαν οι τροπολογίες τελική ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ομόφωνα συγχαρητήρια στον εισηγητή και στην ομάδα που τον πλαισιώνει Φτάσαμε στο τέλος των γνωμοδοτήσεων. Όμως, πριν από την μεγάλη συζήτηση για το Brexit, μένει ακόμη το ψήφισμα για τις προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019 που ε, έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη με απόφαση του Προεδρείου μας και για το ψήφισμα αυτό υπάρχει ένας αριθμός αρκετά σημαντικός 38 τροπολογιών. Θα σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι στις παρεμβάσεις σας για να μπορέσουμε να αρχίσουμε εγκαίρως τη συζήτηση για τη Βρετανική αποχώρηση. Ποιο επιθυμεί να λάβει το λόγο για το ψήφισμα καθεαυτό. No. Όχι, φαίνεται ότι κανείς δεν θέλει το λόγο. Θέλετε το λόγο? Μάλλον όχι κλείνει η συζήτηση και φτάνουμε στις τροπολογίες. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Le vote est clôturé et Πέρας, εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία 3 και καταπέπτει 4 και 5 αν εγκριθεί. Υπέρ της 3 κατά εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψήφος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Le vote est clôturé. Πέρας. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 15 υπέρ κατά απορρίπτεται 16 υπέρ κατά εγκρίνεται 17 υπέρ κατά εγκρίνεται 18 υπέρ κατά εγκρίνεται 19 υπέρ κατά εγκρίνεται 20 υπέρ κατά εγκρίνεται 21 υπέρ κατά επαληθεύουμε ηλεκτρονικά Le vote est clôturé et l'amendement Πέρας εγκρίνεται η τροπολογία. 22. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται 26 υπέρ κατά εγκρίνεται 27 υπέρ κατά εγκρίνεται 28 υπέρ κατά εγκρίνεται 29 υπέρ κατά απορρίπτεται 30 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 31. Για την 31. να έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που προείπα. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτής της τροπολογίας η οποία κάνει λόγο για την προσχώρηση στη σύμβαση του Μαρακές Ορισμένα κράτη-μέλη ήδη ε, έχουν ε, λάβει απόφαση σε σχέση με το σύμφωνο του Μαρακές, μερικοί το έχουν προσυπογράψει, όμως πολλά κράτη-μέλη δεν κύρωσαν τη σύμβαση του Μαρακές. Και ορισμένα κράτη-μέλη σαν το δικό μου δεν έχουν ακόμα αποφασίσει. Αναρωτιέμαι λοιπόν κατά πόσο αυτή θα είναι μια πολύπλευρη προσέγγιση στη μετανάστευση. Δεν ε, συζητήσαμε για αυτό το σύμφωνο. Ας δούμε τις διαφορές που υπάρχουν ε, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το σύμφωνο του Μαρακές και να δούμε και τις διαφορές μεταξύ περιφερειών. Γι' αυτό θα ήθελα να μην την υποστηρίξετε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι εγκρίνοντας αυτή την τροπολογία, αν αυτό κάνουμε, τότε θα είμαστε συνεπείς με αυτό που συνέβη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε σχέση δηλαδή με προγενέστερες γνωμοδοτήσεις που ενέκρινε η Επιτροπή Περιφερειών, έκθεση Μπόσμαν για παράδειγμα. Άρα συμβαδίζουμε με τα προγενέστερα άλλοι που θα ήθελαν το λόγο. Δεν βλέπω. Περνάμε στην ψηφοφορία. Υπέρ της 31 παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά, εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 36 υπέρ, κατά, επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Le vote est clôturé et l'amendement... Πέρας, εγκρίνεται η τροπολογία. 37. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται και 38 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το τελικό κείμενο. Ποιος είναι υπέρ του ψηφίσματος. Κατά αποχές εγκρίνεται το ψήφισμα με μεγάλη πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πολύ και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας σε λίγα λεπτά.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 Αγαπητέ κύριε Μπαρνιέ, σας ευχαριστούμε πολύ που για μία ακόμη φορά δεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Πριν από δύο χρόνια μας παρουσιάσετε τον οδικό χάρτη όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις εδώ, στην Ολομελιά μας. Φέρατε εις πέρας με ιδιαίτερο ταλέντο την αποστολή σας, το είπατε κι εσείς, πέρα από το δύσκολο αυτό διαζύγιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου να γίνει με τρόπο συντεταγμένο, ομαλό υπέρ των πολιτών, υπέρ τη οικονομική και κοινωνική σταθερότητα, υπέρ μια θετική μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τότε που είχαμε τα αποτελέσματα στο δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών συνέχισε να συνομιλεί με τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ του Ηνωμένου Βασιλείου, διατηρώντα επίση ένα σύστημα διαβούλευση όσον αφορά τι επιπτώσει που θα μπορούσε να έχει το Brexit στο σύνολο των περιφερειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι οι επιπτώσει αυτέ ενδεχομένω να είναι ασυμμετρικέ, όχι μόνο όσον αφορά τον τομέα τη οικονομία, αλλά και όσον αφορά τι πιο εκτεθειμένε τελικά περιφέρειε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών τους τελευταίους 17 μήνες ενέκρινε γνωμοδοτήσεις για το ζήτημα αυτό, αλλά είχε και επαφές επιτόπου Βούλησή μα ήταν οι βασικέ τοπικέ και περιφερειακέ ανησυχίε να ληφθούν υπόψη στην όλη διαδικασία. Οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ τη Ευρώπη των 27 έχουν κάθε συμφέρον το Ηνωμένο Βασίλειο να μπορεί να συνεχίσει να συμμετέχει και πέρα από τη μαυρατική περίοδο σε κάποια κοινοτικά προγράμματα στο τομέα του πολιτισμού, τη εκπαίδευση, τη έρευνα ή ακόμα και τη καινοτομία. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η λύση του backstop, του μηχανισμού ασφάλειας, θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε τις συμφωνίες του Μπέλφαστ και να αποφύγουμε σκληρά άκαμπτα σύνορα μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας και κατά αυτόν τον τρόπο θέλουμε να αποφύγουμε να τεθεί ένα αμφιβόλο η ειρήνη η οποία επετεύχθη με τόσες προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περιφέρειες και οι πόλεις των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουν και προετοιμάζονται για τον Brexit τόσο στην Ιρλανδία, όπου η κατάσταση είναι πιο δεινή, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχουμε, όπως ξέρετε, περιφέρειες ε, οι οποίες ε, βασίζονταν πάρα πολύ για την οικονομική τους ανάπτυξη στις οικονομικές σχέσεις, στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς με το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, να καταφέρουμε να πλησιώσουμε και να συνοδεύσουμε τις πιο εκτεθειμένες περιφέρειες. Σας παρακαλώ πολύ, το μήνυμα αυτό πρέπει να πάει στο Συμβούλιο. Πρέπει να καταλάβετε ποιε είναι οι ανησυχίε που έχουμε όσον αφορά την μελλοντική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου. Χαίρομαι πάρα πολύ που στην πολιτική δήλωση κάνετε αναφορά στον πολιτικό διάλογο, ο οποίο σε όλα τα επίπεδα, λέτε, θα πρέπει να αναπτυχθεί, προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή διακυβέρνηση των μελλοντικών μα σχέσεων. Και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν, ότι υπάρχουν και πολλά περιφερειακά κοινοβούλια, τα οποία θα εμπλακούν στην ακύρωση τη μελλοντική συμφωνία αποχώρηση. Κύριε Μπαρνιέ, το Brexit δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θέλουμε, είμαστε πάρα πολλές περιφέρειες, τοπικές και περιφερειακές αρχές που θέλουμε να φέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη. Από κοινού λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα κοινό χώρο ειρήνης και ευημερία. Κύριε Μπαρνιέ, με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα τώρα να σας δώσω το λόγο. Mesdames et les Président, Κυρίες ε, και κύριοι Υπουργοί, Δήμαρχοι, απευθύνομαι σε όλους εσάς ε, που είστε μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και που σας γνωρίζω πολύ καλά. Πρόεδρε Καρλ Χάιντς, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβρίσκω εδώ και που μπορούμε να συνεχίσουμε το διάλογο που ήδη ξεκινήσαμε στο παρελθόν όσον αφορά το Brexit στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Σας είχα ενημερώσει και για τα προηγούμενα στάδια της διαδικασίας αυτής και στις προηγούμενες, στα προηγούμενα καθήκοντα που είχα, προτού γίνω διαπραγματευτής, ήμουνα πάντα σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Ήμουνα και εγώ επικεφαλής μιας περιφέρειας της Γαλλικές Άλπης, στη Σαββοία, στη Γαλλία, Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι στα πλαίσια των νέων καθηκόντων μου, ως επικεφαλής διαπραγμάτευσης δηλαδή για τον Brexit, αλλά και ως Ευρωπαίος Επίτροπος στο παρελθόν, αυτό το οποίο έμαθα ερχόμενο σε επαφή με τους τοπικά ερετούς, με τους επιχειρηματίες, με τους τοπικούς και περιφερειακούς συλλόγους, είναι ζητήματα τα οποία εμπλούτησαν πάρα πολύ το έργο μου και ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα για μένα. Συνεχίζω λοιπόν το διάλογο αυτό και δεν ξεχνάω ποτέ, κύριε Πρόεδρε, ότι την τελευταία φορά που ήρθα εδώ και μου το θυμήσατε τότε, στις 22 Μαρτίου συγκεκριμένα 2017, επτά ημέρες προτού η Τερέζα Μέη απευθύνει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση την επίσημη επιστολή κοινοποίηση της πρόθεσης αποχώρησης μετά το δημοψήφισμα για το Brexit, επιστολή η οποία κινητοποίησε την όλη διαδικασία Μάρτιος 2017 λοιπόν και τώρα έχουμε φτάσει, φτάσαμε μέχρι το Μάρτιο θα φτάσουμε μάλλον μέχρι το Μάρτιο του 2019, την ημερομηνία δηλαδή εκείνη κατά την οποία επίσημα το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξαναβρήκα το λόγο που σας είχα εκφωνήσει τότε και τον ξαναδιάβασα πρωτού έρθω σήμερα εδώ πέρα, γιατί θεωρώ ότι είναι πάντα πολύ σημαντικό να ελέγχει και να επαληθεύει κανείς αν τα όσα λέει στο παρελθόν όντω ισχύουν και είναι ορθά. Σας είχα πει τότε κάτι το οποίο πιστεύω ότι εξακολουθεί και είναι ορθό, ότι το Brexit είχε, έχει και θα έχει πολλές συνέπειες. Πολύ συχνά συνέπειες τις οποίες υποεκτιμούμε, συνέπειες τις οποίες δεν εξηγούμε σωστά, ανθρώπινες συνέπειες κοινωνικές, τεχνικής και νομικής φύσης, χρηματοπιστωτικής φύσης, οικονομικής φύσης. Σας είχα πει επίσης τότε ότι θα δείχναμε απόλυτη αποφασιστικότητα, τουλάχιστον εγώ, τότε ξεκινούσα, ξέρετε, με τα νέα μου αυτά καθήκοντα, θα έδειχνα και εγώ, αλλά και η ομάδα μου, η διαπραγματευτική, την οποία κατάφερα να συστήσω και με την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του κ. Γιούνκερ, αλλά και με όλε τι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασιζόμενο επίση στην εμπειρογνωμοσύνη των μελών του Συμβουλίου αλλά και των κρατών μελών. Σα είχα πει λοιπόν τότε ότι ήμασταν απόλυτα αποφασισμένοι να καταλήξουμε σε μια συμφωνία συντεταγμένη έφτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι αυτό αξίζει πολύ περισσότερο και είναι πολύ πιο σημαντικό από το να έχουμε μία άτακτη αποχώρηση του Μέντου Βασιλείου. Συζητήσαμε επίσης και για τις προποθέσει επιτυχίας τη διαπραγμάτευσης αυτή, Όχι κατά των Βρετανών σε καμία περίπτωση, αλλά μαζί με τους Βρετανούς, στο πλευρό τους. Οι προποθέσει αυτές ήταν ότι θα έπρεπε να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε την ενότητα των 27 κρατών μελών μέσω διαλόγου και διαφάνεια, ότι θα έπρεπε να ανταποκριθούμε το συντομότερο δυνατό στις διάφορες ε, αβεβαιότητες που θα δημιουργούσε η πρόθεση του Μένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές αβεβαιότητες για πάρα πολλούς παράγοντες και είχα πει τότε ότι θα έπρεπε να βάλουμε μια τάξη στα πράγματα. Δηλαδή, καταρχάς να δούμε πώς θα διεξαχθεί το διαζύγιο αυτό, διαχωρισμός ή αποχώρηση, αν θέλετε, και πώς στη συνέχεια θα διαμορφωθεί η μελλοντική σχέση, η μελλοντική εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Διατηρήσαμε λοιπόν την μέθοδο αυτή τότε που σας παρουσίασα και νομίζω ότι πραγματικά ανταποκρίθηκα στις υποσχέσεις που σας δόθηκα τότε. Έκτοτε πήγα δύο με τρεις φορές σε κάθε ένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συναντήσω σε κάθε περίπτωση τους πρωθυπουργού, την κυβέρνηση, τα κοινοβούλια, Συνδικαλιστικέ οργανώσει του εκπροσώπου των επιχειρηματιών. Είχα επίση τη δυνατότητα να πάω σε πολλέ περιφέρειε. Πήγα στη Δανία, την Ιρλανδία, στη Φλάνδρα, στην Κάτω Σαξονία και σε άλλε περιφέρειε. Είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα πνεύμα ενότητα εδώ στι Βρυξέλλε, στο πλαίσιο τη συνεργασία που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεργασία με την, τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των εκατοντάδων αυτών συναντήσεων που είχαμε και με την πολύ στενή συνεργασία που είχαμε και εδώ, στο κτίριο αυτό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώ επίση και με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να λοιπόν πώ καταφέραμε στην πράξη και ίσω για πρώτη φορά στα πλαίσια μια τόσο σοβαρή και πολύπλοκη διαπραγμάτευση, να λοιπόν πώ καταφέραμε να κάνουμε αυτό το οποίο αποκαλώ co-building, δηλαδή μια από κοινού οικοδόμηση του σχεδίου αυτού αποχώρησης με την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν οι ευρωβουλευτές και οι εκπρόσωποι των κρατών μελών. Ξέρω κύριε Πρόεδρε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ανέκαθεν γνώριζε ότι υπήρχε ανάγκη για ενότητα και ότι υπήρχαν συγκεκριμένες προποθέσει για την ενότητα αυτή. Διαφάνεια, Δημόσιο διάλογο, προποθέσει που επιτρέπουν στον καθένα να παίρνει το λόγο, να εκφράζεται, να εκφράζει ανησυχίε και τι ε, τοπικέ ιδιαίτερότητε. Επίσης εδώ στις Βρυξέλλες ε, ήρθα σε επαφή με όσους το ζήτησαν, με πολλούς εκπροσώπους περιφερειών, με προέδρους από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, τις οποίες δεν ξεχνάω ποτέ, και αφουγκράστηκα και τις δικές τους ανησυχίες. Και να λοιπόν πώς, και αυτό ήταν ο ρόλος μάλωστε, να λοιπόν πώς καταλήξαμε σε μια κοινή γραμμή, να πώς καταλήξαμε σε κάποιες κοινέ προτεραιότητες, ε, τις οποίες εκφράσαμε κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν. Τώρα, στη συνθήκη για την αποχώρηση για τον Brexit που το βλέπετε εδώ πέρα, 600 σελίδες, σας καλώ να τις μελετήσετε. Μόλον ότι ενδεχομένω το κείμενο είναι κάπως πολύπλοκο και ενδεχομένω να πέσει βαριά η μελέτη αυτή κατά τη διάρκεια των χρωστινιάτικων διακοπών. Παρ' όλα αυτά, στο κείμενο αυτό προσπαθήσαμε να απαντήσουμε με κάθε δυνατή ακρίβεια σε όλες τις αβεβαιότητες και τις ανησυχίε που δημιουργεί το Brexit. Και γι' αυτό ακριβώς το κείμενο αυτό είναι πυκνό είναι μια συνθήκη, δεν είναι ένας απλός λόγος, μια απλή παρουσίαση. Είναι ένα νομικό κείμενο το οποίο θα πρέπει να δημιουργήσει ασφάλεια δικαίου εκεί που δημιουργεί νομική αβεβαιότητα το Brexit. Καταρχάς για τους πολίτες. 4,5 εκατομμύρια πολίτες 3,5 εκατομμύρια από τα 27 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ζουν και εργάζονται στο Μένο Βασίλειο και από την άλλη πλευρά 1,5 εκατομμύριο Βρετανοί πολίτε οι οποίοι ζουν και εργάζονται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις δικές σας τις περιφέρειες. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δώσουμε απαντήσεις και μια κάποια βεβαιότητα, ασφάλεια δικαίου εκεί που είχε δημιουργήσει η αβεβαιότητα το Brexit. Και θα αναφερθώ λίγο αργότερα επίση και στον δημοσιονομικό κανονισμό. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών διαπραγματεύσεων πάντως προσπαθήσαμε να επιβεβαιώσουμε και ποτέ με επιθετικότητα, το τονίζω αυτό, ποτέ με διάθεση εκδίκηση ή τιμωρία. Αυτό αντιτίθεται πάρα πολύ στα πιστεύω μου. Προσπαθήσαμε να προωθήσουμε τι αρχέ μα, τι οποίε γνωρίζουν πολύ καλά οι Βρετανοί, γιατί ε, από κοινού θέσαμε εδώ και 44 χρόνια τα θεμέλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο και αναφέρομαι εδώ στην ακαιρεότητα της εσωτερικής ενιαίας αγοράς, στο, την αδιέρετες οι τέσσερις ελευθερίες και στην αυτονομία λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Και καταλήξαμε λοιπόν στην συμφωνία αυτή που εγκρίθηκε από τους 27 αρχικούς κρατών και κυβερνήσεων την προηγούμενη εβδομάδα με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και με την υποστήριξη της κυβέρνησης του Μένου Βασιλείου. Πρόκειται για μια συμφωνία αποχώρησης ισορροπημένη η οποία, οφείλω να το πω, και το λέω αυτό με ηρεμία αλλά και με σοβαρότητα, είναι η μόνη και η καλύτερη δυνατή λύση. Η συμφωνία αυτή αποχώρησης δημιουργεί τις δυνατότητες μιας φιλόδοξης μελλοντικής σχέσης άνευ προηγουμένου με το Ηνωμένο Βασιλείο σε πάρα πολλούς τομείς συνεργασίας. Ο πρόεδρο Τούσκα, όπω και ο πρόεδρο Γιούγκερ, υπενθύμησαν ότι είναι πολύ σοβαρή η στιγμή αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε καμία περίπτωση θα πρέπει να γιορτάζουμε, δεν υπάρχει λόγο να γιορτάζουμε και ως διαπραγματευτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σας πω ότι η διαπραγμάτευση αυτή είναι αρνητική, είναι μια αρνητική διαπραγμάτευση. Το Brexit δεν επιφέρει καμία προστιθέμενη αξία για κανέναν. Είναι αμοιβαία δυσμενή, αν θέλετε, η αποχώρηση αυτή και τι δύο πλευρέ. Επομένω, θα πρέπει εμεί να περιορίσουμε τι δεινέ συνέπειε και αυτό ακριβώ προσπαθήσαμε να πετύχουμε μέσω αυτή τη συμφωνία συνθήκη αποχώρηση. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο πιο συγκεκριμένα τώρα σε αυτή την συμφωνία αποχώρηση που έχω ενώπιόν μου. Αναφέρεται καταρχά στι προτεραιότητε των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προηγούνται οι πολίτε, citizens First. Αυτό ήταν το πρώτο μέλημά μας και καταφέραμε να βρούμε μία λύση μαζί με τους Βρετανούς προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και την ασφάλεια των 4,5 εκατομμυρίων αυτών πολιτών καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους να καταφέρουν να διατηρήσουν τα δικαιώματά τους μέχρι το τέλος της μεταβατικής περίοδου. Μετά τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν διαφορετικά. Μετά την επίσημη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και μετά τη λήξη της μεταβατικής περίοδου θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με τους Βρετανούς για το θέμα της κινητικότητας. Δεν θα έχουμε όμως την σημερινή ελευθερία κυκλοφορίας. Πάντως, τα υφιστάμενα δικαιώματα κατοχυρώνονται. Το Brexit, το είπατε και εσείς πριν από λίγο κύριε Πρόεδρε, δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, δεδομένων των προϋποθέσεων ειρήνευσης και σταθερότητας της Συμφωνίας του Μπέλφαστη, της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, αν θέλετε. Εμείς Δεσμευθήκαμε από κοινού με τους Βρετανούς να κάνουμε κάθε τι το δυνατό, our best endeavors είπαμε, προκειμένου πριν από την 1η Ιουλίου του 2020 να εγκρίνουμε και να κυρώσουμε μια συμφωνία εταιρική σχέσης που θα επιλύει και θα διευθετεί τα προβλήματα αυτά. Καθότι όμω δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή βεβαιότητα όσον αφορά την έκβαση των μελλοντικών διαπραγματεύσεων και δεδομένων τη κοινή δέσμευση που έχουμε μαζί με του Βρετανού να αποφύγουμε σε κάθε περίπτωση άκαμπτα σκληρά σύνορα μεταξύ Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία, συμφωνήσαμε για αυτό το οποίο ονομάζουμε backstop, μηχανισμό ασφάλεια. Μία εγγύηση ουσιαστικά, ένα εχέγγυο το οποίο θα είναι νομικά δεσμευτικό, λειτουργικό και το οποίο θα αποτρέψει την επιστροφή άκαμπτων συνόρων στην ίσο της Ιρλανδίας και θα επιτρέψει μια ομαλή συνεργασία μεταξύ του βόρειου και του νότιου τμήματος της νήσου, ιδίως όσον αφορά την εσωτερική αγορά. Θα προσπαθήσουμε να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το backstop, δηλαδή θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία προκειμένου να μην έχουμε σύνορα μεταξύ των δύο περιοχών της Ιρλανδίας, αλλά υπάρχει το backstop ως ίστατη λύση, ως μια εγγύηση, ως παράγοντας σταθερότητας και εγγράφεται ουσιαστικά στην συνέχιση της διαδικασίας ειρήνευσης προς το συμφέρον του συνόλου της Ιρλανδίας, όπως άλλωστε λένε όλοι οι πολίτες, οι επιχειρηματίες και άλλοι παράγοντες και από τη Βόρεια Ιρλανδία. Ένα άλλο σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εσά είναι το ζήτημα του προπολογισμού. Όπως ξέρετε, έχουμε δεσμευτεί, δεσμευόμαστε μάλλον κάθε, 7 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση των πολιτικών μας. Σήμερα το πρωί ουσιαστικά συζητήσατε και τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Το 2014 λοιπόν 28 κράτη-μέλη με τη συνεργασία του Μένου Βασιλείου αποφασίσαμε για τις πολιτικές που θα ακολουθήσουμε και για τη χρηματοδότησή τους μέχρι τα τέλη του 2020. Καταφέραμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι ό,τι αποφασίστηκε με τους 28 θα χρηματοδοτείται και από τους 28 και όχι μόνο από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πέρασε στη συμφωνία και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει απέναντι στις περιφέρειες της πόλης όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική, όσον αφορά τη συνεργασία των πανεπιστημίων, όσον αφορά την υποστήριξη για τις επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν πλέον αυτή τη συμφωνία αποχώρησης. Προσπαθήσαμε στα πλαίσια τους να δώσουμε απαντήσεις σε αναρρύθμιτα προβλήματα. Οι Βρετανοί φεύγοντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόματα και από νομικής πλευράς εγκαταλείπουν 700 διαφορετικές συμφωνίες. Για παράδειγμα, την κοινή αγορά, την Ευρατόμα, τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, πολλές διεθνείς συνθήκες. Όλα αυτά είναι άμεση συνέπεια του Brexit. Αλλά έχουμε και άλλα προβλήματα, όπως για παράδειγμα η προστασία των εμπορικών σημάτων. Ένα εκατομμύριο εμπορικά σήματα τα οποία προστατεύονται από τον οργανισμό που έχουμε στο Αλικάντε της Ισπανίας και γι' αυτό το ζήτημα έχουμε μια συμφωνία προκειμένου να καταφέρουμε να προστατεύσουμε το 1 εκατομμύριο εμπορικά σήματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε επίσης να προστατεύσουμε 3.000 γεωγραφικές ενδείξεις προέλευσης όσον αφορά το τυρί, όσον αφορά τον ίνο, το ελαιόλαδο, που ξέρετε ότι είναι προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την οικονομική ανάπτυξη πολλών περιφερειών όπως για παράδειγμα το ουίσκι, η παρμεζάνα, το σκοτσέζικο ουίσκι, σας δίνω κάποια παραδείγματα. Καταλήξαμε σε μια συμφωνία όσον αφορά μια μεταβατική περίοδο που ζήτησε η Βρετανική κυβέρνηση, μεταβατική περίοδος που θα ξεκινήσει αμέσως μετά την αποχώρησή τους, δηλαδή μετά τα τέλη Μαρτίου και που θα, θα κρατήσει 21 μήνες, ενδεχομένως 1-2 χρόνια Επιπλέον, αν το αποφασίσουμε από κοινού, μεταβατική περίοδος κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θα συμμετέχει στο Ελεκτικό Συνέδριο, δεν θα συμμετέχει στην Επιτροπή των Περιφερειών, δεν θα συμμετέχει στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. επιλογή του Ηνωμένου ήταν αυτή. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια των 21 μηνών τη μεταβατική περίοδου θα βρίσκεται στο στερικό τη Τελωνιακή Ένωση Ιστορική Αγορά και θα συμμετέχει σε όλε τι ε, κοινοτικέ πολιτικέ σεβόμενο τις ε, υποχρεώσεις του και έχοντας τέτοια δικαιώματα. Πολύ ε, τηλεγραφικά και γρήγορα αυτά είναι τα βασικότερα στοιχεία αυτής της συνθήκης αποχώρησης και με τη σύμφωνη γνώμη βέβαια του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αποτελέσει τελικά την τελική συμφωνία αποχώρησης. Τώρα, για μένα, πέρα από το διαζύγιο, πέρα από τον διαχωρισμό αυτών, πέρα από την αποχώρηση, το πιο σημαντικό είναι το μέλλον. Η σχέση δηλαδή που θα οικοδομήσουμε στο μέλλον με το Ηνωμένο Βασίλειο, με μια χώρα η οποία μολονότι θα βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το αποφάσισε, θα παραμείνει μια φιλική χώρα, μια χώρα εταίρος, μια χώρα σύμμαχος. Θα πρέπει λοιπόν να διαμορφώσουμε με έναν εναλλακτικό τρόπο τη συνεργασία μας, την οικονομική μας εταιρική σχέση, τη συνεργασία για την ασφάλεια, πέρα από αυτά που κάνουμε ή που θα κάνουμε μαζί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, και θα πρέπει να καταφέρουμε να ενισχύσουμε την υφιστάμενη φιλία. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να καταλήξουμε σε μια πολιτική δήλωση, την οποία μπορεί να διαβάσει κανείς πιο εύκολα από τη συνθήκη, είναι μόνο 26 σελίδες, μια πολιτική δήλωση η οποία θέτει το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης με τον Ομένο Βασίλειο. Θα ήθελα εξ αρχής να σας πω την απόλυτη αλήθεια κυρίες και κύριοι. Μετά το Brexit τα πράγματα δεν μπορούν να κινηθούν με το συνήθι τρόπο. Δεν θα έχουμε το λεγόμενο business as usual. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως το παρελθόν. Το Brexit θα έχει συνέπειες και αλλάζει τα δεδομένα. Και όπως το έχω πει πολύ συχνά, η καλύτερη σχέση που μπορεί να έχει κανεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να είναι μέλο της Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν είμαστε μέλο της Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή δεν το θέλουμε ή επειδή θέλουμε να αποχωρήσουμε, αναγκαστικά βρισκόμαστε σε μια διαφορετική, λιγότερο ευνοϊκή θέση. Πάντω, το κοινό αμοιβαίο συμφέρον μα είναι να έχουμε μια φιλόδοξη εταιρική σχέση και ακριβώ αυτό περιγράφουμε σε αυτή την πολιτική δήλωση. Μια εταιρική σχέση στον οικονομικό τομέα, για τα αγαθά, για τι υπηρεσίε, για το ψηφιακό περιβάλλον, για την κινητικότητα των πολιτών, για τις μεταφορές, για τις δημόσιες αγορές, για την ενέργεια, αλλά και για την εσωτερική ασφάλεια, για την δικαστική και αστυνομική συνεργασία, αλλά και για την εξωτερική πολιτική, την εξωτερική ασφάλεια και την άμυνα. Αυτή η φιλόδοξη εταιρική σχέση, αν το αποφασίσουμε και αν το θέλουμε από κοινού, εμείς είμαστε έτοιμοι πάντως, θα βασίζεται σε μια συνθήκη ελεύθερων συναλλαγών, χωρίς δασμούς και χωρίς ποσοστώσεις για τα αγαθά και με ένα δασμολογικό καθεστώς που θα προβλέπεται στη Συμφωνία Αποχώρησης που θα λειτουργήσει προς το συμφέρον των επιχειρήσεων και από τις δύο πλευρές της μάχης. Επίσης θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια νέα συμφωνία για την αλία γιατί οι Βρετανοί αποχωρούν και από την κοινή αλληλευτική πολιτική. Επομένω, η μελλοντική αυτή αλληλευτική συμφωνία θα πρέπει να, έχει να, κάνει, θα πρέπει να ρυθμίζει μάλλον την, προσχώ, την πρόσβαση στα ύδατα και την πρόσβαση στην ελευτική αγορά και θα αποτελέσει και αυτή αντικείμενο διαπραγμάτευση στα πλαίσια της μελλοντική μας οικονομικής σχέσης. Εμείς έχουμε δεσμευτεί για το σημαντικό αυτό ζήτημα. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά το ζήτημα αυτό, καθότι υπήρξε υπουργό Αλία στη Γαλλία για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε δεσμευτεί, λοιπόν απέντη στο Μένο Βασίλειο να κάνουμε κάθε το δυνατό προκειμένου να εγκριθεί η συμφωνία αυτή πριν την 1η Ιουλίου του 2020, δηλαδή πριν το τέλος της μεταβατικής περίοδου. Τέλος. Η εταιρική αυτή σχέση ανταποκρίνεται σε πολλές ανησυχίες, που έχουν εκφραστεί από τις πόλεις και τις περιφέρειες που εκπροσωπείτε. Κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να διατηρήσουμε τη δυναμικότητα που έχουμε σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και ξέρω ότι υπάρχουν ορισμένε περιφέρειες και πόλεις που από οικονομικής πλευράς αλλά και λόγω εγκύτητας είναι πάρα πολύ στενά δεμένες με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Προφανώς η εσωτερική αγορά αποτελεί το βασικό μας πλεονέκτημα θα πρέπει πάντως να αξιολογήσουμε και τις επιπτώσεις που θα έχει το Brexit σε σχέση με τη φύση της μελλοντική σχέσης που θα έχουμε με το Νομένο Βασίλειο, πιο συγκεκριμένα για συγκεκριμένε περιφέρειες, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις σχέσεις και τους δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί με το Νομένο Βασίλειο. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακριβώ για αυτό το λόγο, λοιπόν, αποφασίσαμε να υπάρχουν συγκεκριμένε υποχρεώσει προκειμένου να έχουμε αυτό το λεγόμενο level playing field σε οικονομικό, φορολογικό, περιβαλλοντικό επίπεδο ή σε επίπεδο κρατικών ενισχύσεων. Η ιδιαιτερότητα των σχέσεων έγκυται στο ότι στις εμπορικές μας σχέσεις με μια τρίτη χώρα δεν θα πρόκειται για μια συμφωνία όπως ισχύει για την Ιαπωνία, την Κορέα ή τον Καναδά για να φτάσουμε σε μια αριθμιστική σύγκληση. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να ρυθμίσουμε τους κινδύνους απόκλησης, έτσι ώστε η απόκληση αυτή να μην οδηγήσει σε dumping κατά ημών. Θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Παράλληλα, θα πρέπει να διατηρήσουμε τη δυνατότητα συνεργασίας που έχετε εσείς με τις πόλεις και τις περιφέρειες ε, της Μεγάλης Βρετανίας και τα πανεπιστήμια τους. Εδώ, ως προς τη Βόρεια Ιρλανδία, θα παγιοποιήσουμε το πρόγραμμα Peace. Εγώ γνώρισα πάρα πολύ καλά αυτό το πρόγραμμα γιατί ήμουνα υπεύθυνο της ε, ε, περιφερειακής πολιτικής μερικά χρόνια πριν και πέρα από αυτό το πρόγραμμα, ορισμένα προγράμματα θα διακοπούν Γι' αυτό οι Βρετανοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προγράμματα της Ένωσης που είναι ανοιχτά σε τρίτες χώρες ως προς την έρευνα και καινοτομία, την νεότητα, το πολιτισμό και την εκπαίδευση με το Εράσμους και την πολιτική ασφάλεια των περιφερειών. Αυτό αφορά και την διαπεριφερειακή συνεργασία μέσω προγράμματος Interreg που ανοίγουμε προς τις τρίτες χώρες κατά τον προσεχή προγραμματισμό. Παράλληλα, το ίδιο θα ισχύσει και με τη συμμετοχή σε άλλα προγράμματα των Βρετανών, αλλά υπό διαφορετικούς ε, χρηματικούς, ε, οικονομικούς και νομικούς όρους από ό,τι σήμερα. Ε, έχουμε ξεκινήσει ένα διάλογο για την έρευνα και την καινοτομία, για παράδειγμα, και οι δικές σας περιφέρειες θα λάβουν τη σκητάλη για να προωθήσετε έναν διάλογο με τις ε, περιφέρειες της Μεγάλης Βρετανίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Απλώς να υπενθυμίσω ότι εάν επιτύχουμε με κοινή θέληση, αυτή η εταιρική σχέση θα είναι χωρίς προηγούμενο. Αν λάβουμε υπόψη το εύρος και τον αριθμό των ε, πρωτοβουλειών και των ρυθμίσεων που θα δώσουν την πρέπουσα θέση και στις περιφέρειες. Τα περιφερειακά κοινοβούλια θα έχουν το λόγο ένα σημαντικό πολιτικό ζήτημα ως προς το μέλλον έχει ως εξής. Πέρα από την κύρωση του Brexit από εμάς και τη Μεγάλη Βρετανία, οι μελλοντικές σχέσεις θα βασίζονται σε μικτές συμφωνίες με διαφορετική νομική βάση απαιτώντας ε, την ε, ομόφωνη κύρωση από τα 27 Εθνικά Κοινοβούλια και τα περιφερειακά, εκεί όπου χρειάζεται. Δεν βρισκόμαστε στο τέλος αυτού του δρόμου που είναι μακρύς και δύσβατος, αλλά είμαστε έτοιμοι για να οικοδομήσουμε αυτή την εταιρική σχέση όλα αυτά υπό τον όρο ότι θα κυρωθεί αυτή η συνθήκη που είναι η βάση όλων. Εάν δεν κυρωθεί δεν υπάρχει ούτε μεταβατική περίοδος ούτε οικοδόμηση εμπιστοσύνης που χρειαζόμαστε για να χτίσουμε τις σχέσεις μας στο μέλλον. Χρειάζεται κύρωση και από τις δύο πλευρές, και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Βρετανικό βεβαίως. Τώρα ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Ξέρετε ότι οι Βρετανοί θα αποφανθούν επί του κειμένου και των μελλοντικών σχέσεων τις προσεχείς ημέρες για να δεσμευτούν μελλοντικά και εμείς θα τηρήσουμε τις ε, προθεσμίες του δημοκρατικού διαλόγου με τη Μεγάλη Βρετανία από πλευράς ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις 22 Μαρτίου ενώπιον σας μίλησα για τις ε, προκλήσεις και τη νέα ευρωπαϊκή ατζέντα, η οποία δεν συνοψίζεται μόνο στο Brexit. Στην επιστολή κοινοποίησης στο Ηνωμένο Βασίλειο Έκτοτε δηλαδή η Επιτροπή του Jean-Claude Juncker υπέβαλε πληθώρα προτάσεων σε πολλούς ε, τομείς. Μιλάμε για την ενότητα των Ευρωπαίων σε αυτή τη ε, διαπραγμάτευση η θελημένη από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων γιατί πρόκειται για μια σοβαρή κατάσταση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη σοβαρότητα του εγχειρήματος δηλαδή τι θα συμβεί στο βορρά, στο νότο, στη Μεσόγειο, τι θα γίνει ως προς την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ποιες θα είναι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ. Αυτό διαισθάνθηκα από το διάλογο με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Εγώ και η ομάδα μου ε, έχουμε καλλιεργήσει αυτή την ενότητα με το διάλογο και τη διαφάνεια. Θα ήθελα η ενότητα αυτή που μας διακατέχει σε μία τόσο δύσκολη και αρνητική, και αρνητική διαπραγμάτευση να χρησιμοποιηθεί σε μία θετική ατζέντα για να συμφιλιώσουμε τους πολίτες με την Ευρώπη και να απαντήσουμε σε θέματα κυριαρχίας και γειτονίας που διέπουν την ευρωπαϊκή συζήτηση για την οικονομία, την άμυνα, την διαχείριση του μεταναστευτικού, την εταιρική σχέση με την Αφρική και την Πράσινη Ευρώπη. Είναι πολλά τα ζητήματα που διέπουν μια θετική ατζέντα και ελπίζω η ενότητα που ε, δείξαμε μέχρι τώρα να συνεχίσει να τρέφει αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις και μια θετική ε, ατζέντα που θα είναι υπέρ και των περιφερειών μας. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Μπαρνιέ για την ανάπτυξη του θέματος και πλήρη και σύντομη. Βεβαίως ενός εγγράφου το οποίο ασφαλώς και θα εγγραφεί στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και αν δεν μπορούμε ακόμη να γνωρίζουμε κατά ποιον τίτλο. Ζούμε στιγμές δύσκολες, ωστόσο το μήνυμά σας είναι ταυτόχρονα ένα μήνυμα στραμμένο στο μέλλον. Τα όσα μας είπατε προκαλούν ήδη έντονο ενδιαφέρον των μελών της συνελευσής μας. Ένα δέκατο των μελών μας ήδη έχουν εγγραφεί για να λάβουν τον λόγο. Κάτι που δείχνει βέβαια το έντονο ενδιαφέρον τους. Θα παρακαλέσω τώρα, θα προσκαλέσω όλες και όλους να είστε σύντομοι. Γνωρίζετε τους χρόνους αγορεύσεως, με έχετε άλλωστε εκλέξει ως πρόεδρο για να φροντίζω να γίνονται σεβαστά τα όρια αυτά. Έχω μια μικρή πρόταση. Προχωρήστε αμέσως στην ουσία. Έχω ήδη ευχαριστήσει τον κύριο Μπαρνιέ για τα όσα έπραξε. Νομίζω ότι πραγματικά αξίζει θαυμασμού η εργασία του. Αν όμως ο καθένας από μας περάσει τώρα την μισή ώρα της αγορεύσεώ του για να πει ευχαριστώ και συγχαρητήρια, νομίζω δεν εξυπηρετεί ιδιαίτερα τον στόχο να γίνει η συζήτηση. Καλύτερα να τοποθετηθείτε επί τη ουσία. Πρόκειται για συζήτηση επίκαιρου θέματος, όπως άλλωστε έχουμε συνηθίσει να κάνουμε. Θα δώσω λοιπόν τον λόγο πρώτα στον συνάδελφό μας που πρότεινε την, ε, ε συζήτηση, να γίνει η συζήτηση αυτή, την συνάδελφό μας Birgit Χόνιγκ. Κύριε Μπαρνιέ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Τα θέματα αυτά ομολογώ ότι τα έχετε πάντοτε θέσει ενώπιόν μας και μας έχετε πάντοτε ενημερώσει. Και σας ευχαριστώ για τον Ηράκλειο άθλο που επιτύχατε, ακόμη και αν το αποτέλεσμα δηλαδή ότι θα αποχωρήσει η ε, Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι θλιβερό για όλες και όλου μας, ωστόσο η διαπραγματευτική σας ε, τακτική φάνηκε ότι δεν είχε κάνει εναλλακτική επιλογή. Είναι γεγονός η Βρετανική αποχωρήση, είτε μα αρέσει είτε όχι. Στις 25 Νοεμβρίου θα πρέπει, ή, ε, μάλλον η, η απόφαση της 25 Νοεμβρίου θα πρέπει οπωσδήποτε να ισχύσει ώστε να μην έχουμε από τον Μάρτιο του 2019 μια χαόδη κατάσταση. Όλοι χρειαζόμαστε τη μεταβατική περίοδο και τη διαμόρφωση των μελλοντικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Η δική μου ε, εκλογική περιφέρεια, δηλαδή η κάτω Σαξονία, έχει ιδιαίτερε συνδέσει με, με τη Μεγάλη Βρετανία. Πολλοί Βρετανοί ζουν παροιμήν και εργάζονται. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι άλλωστε και σημαντικός εμπορικός εταίρος, ιδίως για την αυτοκινητοβιομηχανία και τα γεωργικά προϊόντα. Το Brexit λοιπόν για μας έχει πάρα πολύ πικρή γεύση. Παρ' όλα αυτά είμαστε προετοιμασμένες και προετοιμασμένοι. Οι επιχειρήσεις της κατοξαξονίας έχουν ήδη αρχίσει να οργανώνονται ώστε να αναπροσανατολίσουν τις εμπορικές ροές τους. Το 2016 ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο ο δεύτερο εταίρο μα. Τώρα έχει πέσει στην τρίτη θέση ήδη. Ω ε, κυβέρνηση Ομοσπονδιακού Κρατηδίου ενημερώνουμε τους πολίτες μας ήδη από καιρό για τις συνέπειες και έχουμε και στραγγυλή τράπεζα του Υπουργείου μου όπου συνεκρίθησαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς για να ενημερώσουν, να ενημερωθούν και να ενημερώσουν. Και μέσω του διαδικτύου τηρούμε όλον τον κόσμο ενήμερο. Από την νομοθετική άποψη Έχουμε έτοιμο νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο της, ε, του Ομόσπονδου Κρατηρίου μας. Υπάρχει ανάγκη νομικής ασφάλειας για ένα Brexit ε, το οποίο να είναι τακτικό, να μην είναι άτακτο δηλαδή. Έχουμε τα σχέδια λοιπόν αυτά ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε το ταχύτερο δυνατό τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ για τα όσα είπατε για την αλία οι αλληλείς μας πλήττονται ιδιαίτερα από το Brexit διότι δεν, δεν θα επιτρέπεται πλέον να αλλιεύουν ε, μπροστά από τις Βρετανικές ακτές. Μέχρι τον Ιούλιο του 2020 θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία για τα δικαιώματα προσβάσεως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για όλους τους αλληλείς της Βόρειας Θάλασσας και ιδίω βέβαια για την δική μας περιοχή της Κάτω Σαξονίας να μην παραιτηθεί από την προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γνωρίζω, κύριε Παρνιέ, ότι συμπαρατάσσεστε μαζί μα. Αγαπητέ κυρίε και κύριοι, το Brexit θα επιφέρει μεγάλε αλλαγέ σε όλη την Ευρώπη. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις αρχέ και στι αξίε τη και να τι επεκτείνουμε ακόμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο συνάδελφό Μάικλ Μέρφυ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε ανεξαρτήτως των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και έχουμε ακόμη μπροστά μας, χαίρομαι για το σχέδιο συμφωνίας που περιλαμβάνει συμβασμούς και από όλες τις πλευρές και ιδίω από την Ιρλανδική πλευρά η προστασία της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής σε όλα τα τμήματά της. Εγγυάται ότι δεν θα υπάρξει σκληρό σύνορο στο νησί της Ιρλανδίας η ανδήποτε περίσταση. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το σχέδιο πρωτοκόλλου καθιστά απόλυτα σαφές ότι δεν υπάρχει τίποτε στο σχέδιο συμφωνίας το οποίο να θέτει σε κίνδυνο με ενδίποτε τρόπο το συνταγματικό καθεστώς της Βόρειας Ιρλανδίας καθώς επίσης και την αρχή της συνένεσης που περιλαμβάνεται στην Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Η κύρωση του σχεδίου συμφωνίας είναι ο μόνος και ρεαλιστικά ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί μια τακτική βρετανική αποχώρηση που είναι προς το συμφέρον όλων των πόλεων και περιφερειών μας οι οποίες θα πρέπει να συνεχίσουν να προετοιμάζονται. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί. Θα υπάρξουν αλλαγές βαθιές. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιας κλίμακος. Είναι σημαντικό πόλεις, κοινότητες και περιφέρειες να είναι έτοιμες για τις αλλαγές αυτές. Και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Οι περιφέρειες θα πρέπει να είναι οι βασικοί φορείς που θα προετοιμάσουν την ανταπόκριση της αλλαγές αυτές. Επομένως, η Επιτροπή Περιφερειών πρέπει να παραμείνει στον κεντρικό ρόλο μέσα στον διάλογο αυτό που συνεχίζεται για τη Βρετανική αποχώρηση. Υποστηρίζω τους Βρετανούς συναδέλφους μου που ζητούν στενή συνεργασία μετά το Brexit μεταξύ ημών και του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίω ό,τι αφορά το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Ο είναι ο Thank you, President. Ευχαριστώ. Με το Ηνωμένο Βασίλειο κοντά στο συνταγματικό χαός και επειδή την επόμενη εβδομάδα υπάρχει και προοπτική απόρριψης του Brexit και ενός νέου ε, δημοψηφίσματος θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν θα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να μην υπάρξει συμφωνία. Η Ευρώπη των 27 θα μπορούσε να σκεφτεί την επέκταση του άρθρου 50 μετά το Μάρτιο του 19 ή θα ενθαρρύνεται το Ηνωμένο Βασίλειο να αποσύρει το άρθρο 50 όπως όρισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εγώ διαμένω στο Μπέρμιγχαμ, το οποίο ευεργετήθηκε ιδιαίτερα από το, την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να συνεισφέρουμε περαιτέρω. Το Δημοτικό Συμβούλιο μας θέλει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις περιφερειακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κάλφον Λάγκερμαν έχει το λόγο. Η κυρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πολλά ελέγχθησαν για το Brexit και είπατε ότι θα χάσουμε αμοιβαία από αυτή τη συμφωνία. Υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια για το μέλλον. Στην δυτική πλευρά της Σουηδίας εργαζόμαστε στεναρά ε, για το Brexit. Η Handelsbank που είναι μια μεγάλη τράπεζα ετοιμάζεται και για την περίπτωση του Brexit χωρίς συμφωνία. Το μεγαλύτερο λιμάνι, το μεγάλο αυτό λιμάνι, έχει εμπορικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και προσπαθούμε να προβάλλουμε νέα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της αλίας που είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για εμάς. Στα σχολεία, στα λύκεια ε, υπάρχει μια μεγάλη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Αναρωτιέμαι τι θα γίνει για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν και υποτροφίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει να γίνει μία έφτακτη λοιπόν αποχώρηση. Ο κύριος Γιόγκμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό μου προς τον κύριο Μπαρνιέ για το τι κατάφερε. Και αυτό το λέω και εξ ονόματος της ομάδας μου. Πρόκειται για μια φιλόδοξη μελλοντική συνεργασία, όπως είπατε. Μιλάμε για τη συνεργασία τοπικών και περιφερειακών αρχών ε, και συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Πώς διαβλέπετε αυτή τη συνεργασία στο μέλλον. Ο κύριος Μπαρνιέ θα συνεχίσει αυτή την εργασία και μετά το Brexit. Καρλ Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε ε, για μια καλή συμφωνία για ε, να οδηγήσει σε καλές ε, φιλικές σχέσεις. Ένα σκληρό Brexit χωρίς συμφωνία θα οδηγήσει σε ολέθριο αντίκτυπο σε όλες μας τις οικονομίες. Εμείς θα μπορούσαμε να χάσουμε 2,6% του ΑΕΠ και πολλές θέσεις εργασίας και για τις 30.000 κατοίκους ε, υπηκόους της Βρετανίας που ζουν στις Βρυξέλλες καθώς και Βέλγους που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα υπήρχαν σοβαρές συνέπειες. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ετοιμάσουν τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις Χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία ως προς τις ε, κρατικές ενισχύσεις, έτσι ώστε οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να μπορέσουν να δράσουν μακροχρόνια, να δούμε τι θα γίνει στη Βόρειο Θάλασσα, γιατί μιλήσατε για την αλία. Επίσης θα πρέπει να γίνει σοβαρή εργασία στα λιμάνια. Η Φλάνδρα είναι μικρή περιφέρεια, αλλά έχουμε πολύ μεγάλα λιμάνια. Ελπίζω να λάβετε υπόψη τις ιδιαιτερότητες στα κράτη-μέλη. Η κυρία Μπάρμπαρα Άιμπιγκερ. Ομιλώ ως πρόεδρος της Automotive Inc. Πολλά εκατομμύρια εργαζόμενοι εξαρτώνται από την αυτοκινητοβιομηχανία η οποία πλήττεται από το Brexit. Θα σας εξηγήσω για την Steiermark στην Αυστρία όπου η Μεγάλη Βρετανία είναι τέταρτος εταίρος εξαγωγών για, την αυτοκινητοβιομηχανία, όπου υπάρχουν σημαντικές αλυσίδες προμήθειας προς την, προς την ε, ε, Μεγάλη Βρετανία. Για παράδειγμα, το μοντέλο Mini της ε, BMW παράγεται, υποτίθεται, στην Οξφόρδη. Παρ' όλα αυτά, 70% των ανταλλακτικών που αποτελούν το αυτοκίνητο αυτό προέρχονται από ευρωπαϊκή παραγωγή, από αυστριακή παραγωγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξήγαγε το 2017 2,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα στη Μεγάλη Βρετανία. Η αυτοκινητοβιομηχανία λοιπόν θίγεται βαρύτατα από το Brexit και σας παρακαλώ κύριε Μπαρνιέ να το λάβετε ιδιαίτερα υπόψη σας αυτό. Ευχαριστώ. Πέτερ Κάιζερ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, όπως είπε η προλαλήσασα, το Brexit αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Θα πλήξει όλε τι περιφέρειες με διαφορετικό τρόπο και τι κοινότητε. Θα ήταν σημαντικό από τώρα ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το σκεφτεί ότι δηλαδή το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και ιδίω τα κέντρα βάρους περιφερειακής ανάπτυξη αποτελούν ένα τρόπο για να αντιμετωπιστούν οι δυσμενεί αυτέ εξελίξει. Αφετέρου, συγχαρητήρια για, τον, για την ε, συμφωνία εξόδου. Πριν όμω κυρωθεί δεν ισχύει. ποιε προοπτικέ υπάρχουν, ποια προοπτική αναπτύσσετε εσεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν τελικώ αποτύχει. Αν δεν γίνει δεκτή δηλαδή η συμφωνία ε, αποχώρησης. Είναι σημαντικό αυτό για τι χώρε μέλη. Και εν προκειμένου το ερώτημα τι θα γίνει με την φιλόδοξη εταιρική σχέση. Δεύτερο, θα πρέπει να διδαχθούμε ένα πράγμα ως Ευρώπη στο σύνολό μας καθαρά εθνικές σκέψεις και τακτικές οδήγησαν στο να θυγεί αρνητικά ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Φρανσουά Ντεκόστερ. Ευχαριστώ πολύ. Το μήνυμα για το μέλλον είναι η ελπίδα. Ο Πιμπίσερ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Αλίας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσει, κυρία Μπαρνιέ, διότι λάβατε πολύ σοβαρά υπόψη σας την αλία κατά τις διαπραγματεύσεις. Βρισκόμαστε σε ένα ε, σημείο κλειδί μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, διαπραγμάτευσης. Πρόκειται για την εγγύηση της ενότητας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη μέθοδο θα πρέπει να τη διευρύνουμε προς τη διαφάνεια των 27 σήμερα. Θα πρέπει να δείξουμε το ότι να είναι κανείς μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι το ίδιο με το να μη συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και θεματικά. Τι σημαίνει το Brexit για τους που θέλουν να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ξέρουν σε τι συνεισφέρει. Οι μελλοντικές σχέσεις θα πρέπει να είναι θετικές. Έχουμε μεγάλη ανάγκη ως Ευρωπαίοι και ειδικά οι όμορες χώρες ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό αφορά και τους ε, Βρετανούς. Γιατί εγώ δεν θυμώνω με το λαό που υπερψήφισε το Brexit, αλλά ε, θυμώνω με την ανευθυνότητα των πολιτικών ανθρώπων που οδήγησαν σε αυτή την ε, ψήφο. Mr. Barnier, uh, Κύριε Μπαρνιέ, θα ήθελα και εγώ να μιλήσω εξ ονόματος της Σλοβακίας, της χώρας μου και θα ήθελα να πω ότι ανησυχώ με το τι συμβαίνει στη χώρα μου. Οι σημερινές συζητήσεις είναι προσήκουσες γιατί μιλάμε για τις ομάδες αντιευρωπαϊστών που όλο ένα και διονγκώνονται στη χώρα μου. Υπάρχει ένα κόμμα των Ναζί στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο, υπάρχουν ακραίες δυνάμεις, υπάρχουν φιλορωσικές δυνάμεις από τη μία πλευρά και θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και με την Ουκρανία, ποια είναι η στάση των Ρώσων έναντι της Ουκρανίας. Ξέρω ότι θα υπάρχουν συνέπειες και κατά της χώρας μου. Τώρα αποφασίζουμε για το μέλλον της Σλοβακίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επειδή είμαι διοικητής περιφέρειας θα ήθελα να σας ρωτήσω τι πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να αντιστρέψουμε αυτές τις τάσεις και να συστρατευτούμε με την Ευρώπη. Ο Άντωνι Μπιουκάναν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Μπαρνιέ, η ε, Εθνική Ένωση Κόσλα θα ήθελε και το Ηνωμένο Βασίλειο και οι διαπραγματευτές να ξέρετε ποια είναι η προοπτική της Σκοτίας. Εμείς θέλαμε να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρήσαμε ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία για την ευημερία της Σκοτίας αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, μιλήσαμε για την ψήφο του λαού την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή να μπορέσουμε να παραμείνουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε να ανασταλεί το άρθρο 50 μέχρι να γίνει αυτή η ψηφοφορία, η ψηφοφορία και θα θέλαμε την υποστήριξη των Βρυξελών. Αν σταθεί αναγκαίο, θα θέλαμε να υπάρχει ένα κοινό σώμα συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Μάρτιο του 2019 γιατί πολλοί ήταν υπέρ της ε, παραμονής και θα πρέπει οι ε, νόμιμοι εκπρόσωποι των περιφερειών να μπορέσουν να συμμετάσχουν και στις μελλοντικές διαδικασίες. Εάν ε, δεν επιβλέψουμε αυτές τις αλλαγές, αυτό θα σταθεί κατά των Σκοτσέζων που καταψήφισαν το Brexit και θέλαν να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ευγνώμονες. Μετά από τις 12 αυτές ε, παρεμβάσεις θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπαρνιέ για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω όλους όσοι πήραν το λόγο και εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου πολύ γρήγορα, κυρία Μπέργκετ. Αναφερθήκατε πριν από λίγο στην όλη προετοιμασία που γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο. Επικεντρωθήκατε και εσείς αλλά και μια συναδελφό σας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας η Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε 70 ανακοινώσεις ανά τομέα, οι οποίες είναι δημόσιες και οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις αλλά και από τις περιφέρειες, προκειμένου να καταλάβουν καλύτερα τι διακυβεύεται στα πλαίσια της προετοιμασίας, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για το σενάριο το οποίο απευχόμαστε, αυτό του no deal δηλαδή, της μη ύπαρξης συμφωνίας για τον Brexit. Επομένως, οι περιφέρειες σε συνεργασία με τις τοπικές αλλά και εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να αφιερώσουν τον απαραίτητο χρόνο από τώρα μέχρι το Μάρτιο προκειμένου να προετοιμαστείτε. Είναι καλύτερο να επιταχύνετε, αν θέλετε, και τη διαδικασία προετοιμασία. Τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα αν προετοιμαστείτε τώρα από ό,τι αν το αφήσετε μετά. Ο Κάρλο Βαν και ο Πίτερ Κάιζερ Αναφέρθηκαν επίσης στα όλα μέτρα πλησίωσης των περιφερειών. Ο Μάικλ Γκάβιν επίσης αναφέρθηκε σε αυτό. Στην αρχική μου παρέμβαση είπα ότι η πρώτη επίσκεψη που έκανε ήταν στη Φλάνδρα, στην Μπρούζ συγκεκριμένα και είδα εκεί τις δυνάμει επιπτώσεις που μπορεί να έχει το Brexit και το πόσο σημαντικό είναι να καταφέρουμε να συνεχίσουμε τους δεσμούς αυτούς εμπορικούς, δηλαδή εισαγωγέ και Εξαγωγέ περνάνε από ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό λιμάνι. Προκειμένου λοιπόν να παληθεύσουμε πραγματικά, να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις αναπεριφέρεια και να φέρουμε εδώ πέρα στη Δανία, τι Κατοχώρε, το Βέλγιο, στις γαλλικέ επίση περιφέρειε αναφέρομαι, για να αξιολογήσουμε λοιπόν πραγματικά τον αντίκτυπο του Brexit θα πρέπει να γνωρίζουμε την πραγματική φύση των μελλοντικών σχέσεων και να αναφέρω κάτι το οποίο λέγεται και στην πολιτική δήλωση που σας καλώ πραγματικά να διαβάσετε γιατί είναι συγκεκριμένη και πάρα πολύ ανοιχτή και ειλικρινής. Αναφέρεται στις δυνατότητες σύγκλησης. Βάσει των δικών μας αρχών που δεν είναι διαπραγματεύσιμες, ακερότητα της αγοράς, ο ακέρος επίσης χαρακτήρας των τεσσάρων ελευθεριών που δεν μπορούν να διαχωριστούν και από την άλλη αναφερόμαστε επίσης και στη Βρετανική πλευρά. Ο πρόεδρος όμως Συμβουλίου, ο κύριος Τούσκα, του είπε αν κατά τη διάρκεια τη μεταβατική περίοδου μετά τον Brexit που θα κρατήσει δύο χρόνια ενδεχομένω και παραπάνω αν οι Βρετανοί κάνουν άλλα αιτήματα, αν εξελιχθούν αν θέλετε οι απαιτήσει του, εμεί είμαστε σε θέση να προσαρμοστούμε. Η πολιτική δήλωση αναφέρεται στη δυνατότητα σύγκληση για αυτό το οποίο ονομάζουμε Free Trade Agreement ή Free Trade Area, μια συμφωνία, μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Μπορούμε να πετύχουμε κάτι λιγότερο, κάτι και περισσότερο, κάτι ανώτερο πιο αναβαθμισμένο με βάση πάντα τα αιτήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Είμαστε λοιπόν διαλλακτικοί, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι θα διατηρηθούν πάντα ακέρες οι βασικές μας αρχές. Καταγράφω πάντως την ανησυχία που εκφράζουν συγκεκριμένε περιφέρειες. Έχω ήδη συνομιλήσει με τον πρόεδρο Γιούνκερ, με την αρμόδια επίτροπο για τα περιφερειακά κονδύλια. Όταν θα είναι πιο ξεκάθαρο στο μέλλον ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε για την μελλοντική μας σχέση με βάση την ένταση, αν θέλετε, της σχέσης αυτής, πόσο δυνατή ή αδύναμη θα είναι, με βάση τον πραγματικό αντίκτυπο του Brexit, θα καταφέρουμε να αξιολογήσουμε πραγματικά ποιος είναι ο καλύτερος δώσει τρόπος για να πλαισιώσουμε και χρηματοοικονομικά τις περιφέρειες. Η κυρία Καρλαφέγγεν αναφέρθηκε στα πανεπιστήμια. Και για τον Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε τα μέσα και τα εργαλεία αυτά που χρησιμοποιούμε ήδη με τρίτες χώρες όπως το Ισραήλ, η Νορβηγία ή η Ελβετία. Και εκεί συμπεριλαμβάνεται και το πρόγραμμα Εράσμου, το οποίο αναφερθήκατε και εσείς. Στον κύριο Μπόρτερ απευθυνόμενος, λέω ότι καταλαβαίνω απόλυτα τις ανησυχίες του και ο κύριος Μποκανάν αναφέρθηκε στο άρθρο 50 Κύριε Πρόεδρε, αφού γράζομαι πραγματικά τι ανησυχίε σα, αλλά από τη θέση που έχω τώρα του διαπραγματευτή δεν θέλω και δεν μπορώ να εμπλακώ στην συζήτηση που γίνεται σε εσωτερικό επίπεδο στον Εμένο Βασίλειο. Δεν μπορώ, δεν δύναμαι να το κάνω αυτό. Ακούω του πάντε, δέχομαι του πάντε στο γραφείο μου, ακόμα και τον κύριο Φάρατζ. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πρόσφατα μάλιστα μαζί του. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ εγώ άμεσα να εμπλακώ σε αυτή την καθαρά εσωτερική συζήτηση. Γνωρίζετε όλε τι προποθέσει χρησιμοποίηση του άρθρου 50. Κινητοποιήθηκε το άρθρο αυτό από το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν μπορώ εγώ να πω ούτε θα ήθελα να εμπλακώ κάνοντας προβλέψεις για το πώς θα αποφανθεί το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Αυτό που λέω με απόλυτη ειλικρίνεια και ηρεμία μετά από αυτά που είπε και ο πρόεδρος του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συμφωνία αυτή αποχώρησης που έχουμε επιτάπητος και η πολιτική δήλωση αποτελούν για μας τις μόνες και καλύτερες δυνατές λύσεις προκειμένου να έχουμε μια συντεταγμένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και το λέω για μία ακόμη φορά απευθυνόμενο στον κύριο Γιόγκμαν στα πλαίσια της συμφωνία αυτής αλλά και τη πολιτικής δήλωση, υπάρχουν ήδη τα στοιχεία, οι παράμετροι αυτής της ιδιαίτερα φιλόδοξη σχέσης που θέλουμε να έχουμε. Αν ακολουθήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πολιτική δήλωση θα καταλήξουμε σε μία πρωτόγνωρη οικονομική σχέση που δεν έχουμε με καμία άλλη τρίτη χώρα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συναδελφό σα που πήρε τελευταίο το λόγο αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στι ιδιαιτερότητε τη Σκοτία. Προφανώ ασχοληθήκαμε και με τι πτυχέ αυτέ, αλλά ω διαπραγματευτή, εγώ συνομιλώ με την επίσημη κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εδώ και δύο χρόνια μα λέει ότι αποχωρούμε από, την, από το Ηνωμένο Βασίλειο, υπο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποχωρούμε από την Τελωνιακή Ένωση, αποχωρούμε από την εσωτερική αγορά. Πολύ ωραία. Το βρίσκουμε θλιβερό βέβαια αυτό, το καταγράφουμε και το λαμβάνουμε πάντως υπόψη και λέμε ότι θα πρέπει πάντα να ισχύουν βέβαια οι αρχές μας. Ο κύριος Ντρομπά, ο κύριος Κόιστερ και άλλοι προλύσαντες αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις Μάλλον, εγώ αναφέρομαι στις επιπτώσεις του Brexit εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα όμως ήμουνα ερετός, εκπρόσωπος εκλεγμένος από τους πολίτες. Δεν νομίζω λοιπόν θα πρέπει να συγχαίουμε τα διδάγματα στα οποία αναφέρθηκαν οι προαλήσαντες με τις συνέπειες που μπορεί να έχει το Brexit. Ξέρετε ότι στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα στον Ηνωμένο Βασίλειο, όπω και στι ψηφοφορίε που έχουν λάβει χώρα και στι δικέ σα περιφέρειες, εκφράζεται πολλέ φορέ ένα αίσθημα οργή, ένα αίσθημα απομόνωση, το οποίο αισθάνονται οι πολίτε και στο οποίο εμεί θα πρέπει να ανταποκριθούμε θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο ή εθνικό επίπεδο. Οι απαντήσεις υπάρχουν. Πρέπει να ανταποκριθούμε στην οργή όμως αυτή, στο σκεπτικισμό αυτό, αν θέλουμε πραγματικά να αποφύγουμε το λαϊκισμό. Και να προσθέσω κάτι ακόμα κύριε Πρόεδρε, απευθυνόμενο στον κύριο Νταμπράς Ζουράς, ανέκαθεν το έλεγα και εξακολουθώ να το πιστεύω ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε χώρα κάθε εδαφική επικράτεια, κάθε πολίτης αντιστοιχεί σε μια προστιθέμενη αξία. Εσείς αναφερθήκατε στη Σλοβακία. Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιφέρει μια προστιθέμενη αξία σε αυτήν την κοινότητα αξιών που έχουμε δημιουργήσει. Πολύ ωραία. Ας περάσουμε στον δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Ο κύριος Μάρκ Σπάις έχει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όταν είπε το πρώτο όχι η Μεγάλη Βρετανία το 1957, πέρασαν δύο δεκαετίες μέχρι να πει το ναι. Η κάτω Σαξονία δεν θα υπήρχε καν χωρίς τη Μεγάλη Βρετανία. Όμως για να μπορέσει η Μεγάλη Βρετανία να ξαναπεί ναι στην Ευρώπη, πρέπει να διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό ιδεώδες ζωντανό μέσα στην ε, Μεγάλη Βρετανία. Και εδώ αναλαμβάνουν ιδιαίτερη ευθύνη οι περιφέρειες με συναντήσεις, με συνεργασίες στο τοπικό επίπεδο, στο επίπεδο των σχολείων, στο επίπεδο το περιφερειακό, με διαρκή ανταλλαγή. Θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν μπορεί η Βρετανική αποχώρηση να μας οδηγήσει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Αντίθετα, θα πρέπει να τις ενισχύσουμε τις προσπάθειες αυτές. Και επειδή μου μένουν μόνο λίγα δευτερόλεπτα, απευθύνω και πάλι τα ευχαριστή, τις ευχαριστίες μου και τα συγχαρητήριά μου για, την θαυμάσια για τον θαυμάσιο τρόπο με τον οποίο ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων ο κ. Μπαρνιέ. Τώρα ακολουθεί ο κύριος Εθνική Συνέλευση της Ουαλίας. Δεν έχω χρόνο για να αναπτύξω τα αισθήματά μου για την κρίση στην οποία εισερχόμεθα και τις επιπτώσεις του Brexit για τον λαό της Ουαλίας. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μακροπρόθεσε καταστρεφικές συνέπειε, Ό,τι και αν συμβεί πάντως, εμείς οι Ουαλοί θα συνεχίσουμε να θέλουμε να έχουμε μια συνεχιζόμενη ε, επαφή και σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνέλευσή μας. Έχουμε μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων που έρχονται τώρα και οι οποίοι θα συνεχίσουν να θεωρούν τους εαυτού τους ως νεαρούς Ουαλού Ευρωπαίου στο μέλλον. Και ελπίζω σε κάποια στιγμή στο μέλλον να μπορούν να παρακάθεται εδώ, στην παρούσα συνέλευση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποια βήματα μπορούμε να λάβουμε ε, ώστε κοινοβούλια με ε, αποκεντρωμένα όπως το Ουαλικό να μπορέσουν να συνεχίσουν να έχουν σχέσεις και επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες να είναι παραγωγικές και αυτοδύναμες στον κόσμο μετά το Brexit και τι είδους εταιρική σχέση μπορεί να είναι δυνατή ανάμεσα στην Ουαλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να εξασφαλιστεί ότι η φιλία και οι σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει ως τώρα να μπορέσουν να συνεχιστούν, γιατί πρέπει να συνεχιστούν. Ευχαριστώ. Η κυρία Κλαβαγιού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προέρχομαι από την Ισπανία, από μία πόλη με πολλούς αμπελώνες και όπως είπε ο κύριος Βανίρ βρισκόμαστε σε ένα δρόμο γεμάτο αμφιβολίες μέχρι να φτάσουμε στο τελικό σενάριο. Πρόκειται για μία πόλη που εξαρτάται από ένα προϊόν που σχετίζεται με ένα γεωγραφικό προσδιορισμό, δηλαδή το κρασί που χρειάζεται, που χρήζει προστασίες, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ονομασίες προέλευσης που συνδέονται με την ε, τοπική οικονομία. Και τη στιγμή που οι Βρετανοί θα μας ανταγωνιστούν θα πρέπει να προφυλάξουμε τα συμφέροντά μας, να τα διαφυλάξουμε. Θεωρώ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο φεύγει, αλλά δυστυχώς η Ισπανία στο Γιβραλτάρ ε, αντιμετωπίσει μία κατάσταση όπου επικρατούν οι έπικοι. Ε, πρόκειται για έναν ιστορικό αναχρονισμό τον οποίο θα πρέπει να επιλύσουμε. Αυτό πλήττει τους Ισπανούς που εργάζονται στο Γιβραλτάρ και πρέπει καθημερινώς να μεταβαίνουν σε αυτή την πόλη για την εργασία τους. Ο Κορλάμας als burgemeester en bestuurder van de regio ε, Προέρχομαι από το Ρότερνταμ. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης. Προετοιμαζόμαστε για το Brexit και προετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα, ελπίζοντας βέβαια πάντοτε στα καλύτερα. Βλέπουμε και τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία. Προετοιμαζόμαστε, όπως είπα, κάνουμε την προσπάθεια να ενημερώσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις δημιουργούμε βοήθειες για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών του Brexit και έχουμε και ένα Brexit Impact Scan για όλες τις ε, Ολλανδικές περιφέρειες και τοπικές διοικήσεις. Η περιφέρεια του Ρότερνταμ προσπαθεί λοιπόν. Όμως οφείλω να σας πω επίσης ότι η αποχώρηση θα πρέπει για να αντιμετωπιστεί να ε, οδηγήσει και σε επενδύσεις. Είναι σημαντικό να ενισχυθούν, για παράδειγμα, οι λιμενικές εγκαταστάσεις. Πρέπει να προετοιμαστούμε για τον Brexit. Βλέπουμε ότι για τις επιχειρήσεις, παρόλες τις εκκλήσεις, δεν είναι ακόμα καλά προετοιμασμένες. Και για την περιφέρεια του Ρότερνταμ, που είναι το μεγαλύτερο εξαγωγικό και εισαγωγικό λιμάνι, δεν επιτρέπεται να καθυστερήσουμε. Αγαπητέ κύριε Μπανιέ, η ανταλλαγή γνώσεων και η κινητικότητα των νέων είναι από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το δείχνει και η μεγάλη επιτυχία του έρασμος και των ερευνητικών προγραμμάτων γιατί αυτά σημαίνουν όλα βάση συνεργασίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα των επιστημών και της έρευνας είναι κεντρικός εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ιδιαίτερα για την δική μου πόλη, το Βερολίνο. Κατά την επεξεργασία των μελλοντικών σχέσεων συνεργασίας θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια ισορροπία με την έννοια όχι cherry picking όπως λένε στα αγγλικά, αλλά ταυτόχρονα να ανοίξουν οι συνεργασίες η διαίρεση του Βερολίνου, παρόλη τη διαίρεση του Βερολίνου, ε, ε, υπήρξαν συνεργασίες και με την άλλη πλευρά. Η Ιστορία επιτυχία τελικώς, η οποία μπορεί να, χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο και για την Ευρώπη. Η πλήρης αποχώρωση του, της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ερευνητική Κοινότητα θα σημάνει καταστροφή. Δεν χρειαζόμαστε Europe first για να παραφράσω τα λόγια του Αμερικανού Πρόεδρου. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη η οποία να εξασφαλίσει την επιτυχία τη. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπαρνιέ, ως νεότερο μέλος της Ιρλανδικής Αντιπροσωπείας ε, μεγάλωσα σε μια Ιρλανδία όπου επικρατούσε η ειρήνη κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι υποστηρίξατε στεναρά τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και γιατί αναγνωρίσατε τις ολέθριες συνέπειες σκληρών συνόρων μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Ε, όμως, θεωρώ ότι θα πρέπει να προωθήσουμε και συγκεκριμένη δράση στη Βουλή των Κοινοτήτων για να δούμε ποια πορεία θα κρατήσουμε. Εδώ είχαμε προωθήσει ένα ψήφισμα για ένα ταμείο σταθεροποίησης για τις περιφέρειες που θα πληγούν ιδιαίτερα από το Brexit. Θα ήθελα να μας υποστηρίξετε για την δημιουργία αυτού του Ταμείου Σταθεροποίησης. Ευχαριστούμε. Ε, Ανέτ Ταμπαρά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλώ ως πληρεξούσια του Δήμου Αμβούργου που είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική πόλη της ε, Γερμανίας. Έχουμε το τρίτο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό λιμάνι και πάρα πολύ στενές σχέσεις οικονομικές και εμπορικές με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα φυγούμε λοιπόν βαθύτατα από το Brexit αλλά δεν ξέρουμε ακόμη πόσο πολύ. Το καλοκαίρι ξεκινήσαμε με μια ομάδα συντονισμού υπό τη δική μου διεύθυνση, όπου συνέρχονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς, βεβαίως και με εκπροσώπους της ε, οικονομίας, της βιομηχανίας, των κτηνιάτρων και των τελωνιακών υπαλλήλων. Ενημερώνουμε διαρκώς τους πολίτες σχετικά με τις συνέπειες του Brexit και ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε στα συρτάρια μας ένα νομοσχέδιο αφενός για το ενδεχόμενο όπου θα γίνει δεκτή η συμφωνία, αλλά και για το ενδεχόμενο ε, ενός μη συντεταγμένου Brexit. Αυτό που είναι αναγκαίο κατά τη γνώμη μας είναι σε όλα τα επίπεδα, από την Κομισιόν, τα εθνικά ε, κράτη, μέχρι και τις κοινότητες, όλοι να ακολουθούν μία ενιαία γραμμή, διότι η νομοθεσία θα πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα να ακολουθεί την ίδια γραμμή. Χαίρομαι που έχει αρχίσει αυτός ο διάλογος και ευχαριστώ και πάλι τον Μισελ Μπαρνιέ για το θαυμάσιο έργο που έχει επιτύχει. Ακολουθεί ο κύριος Ντρομποσλάβιτ. Les absents ont le prochain... Απόν. Ο κύριος Πασίλο Χόρτα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαρνιέ. Μας ενδιαφέρουν οι μελλοντικές σχέσεις με τη Μεγάλη Βρετανία μετά το Μάρτιο του 2019. Μετά τις 11 Δεκεμβρίου θα δούμε ακριβώς τι θα συμβεί μετά την ψηφοφορία από την Βουλή των Κοινοτήτων. Θα πρέπει να δούμε πώς θα φτάσουμε λοιπόν σε φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εμπορικό εταίρο και φυσικά η Μεγάλη Βρετανία θα παραμείνει μια μεγάλη φίλη. Θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του Brexit και στον τουρισμό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βασιζόμαστε σε ένα 24% σε επίπεδο ε, εισαγωγών που θα πληγούν. Αυτό αφορά και την πόλη μου, την Σύντρα, η οποία η Ρίστο εν παρόδο θα πληγεί ιδιαίτερα από τη μείωση του τουρισμού. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει κατά την μεταβατική περίοδο θα πρέπει να οριστεί σωστά αυτή η μεταβοτική περίοδος. Έχετε υπερβεί το χρόνο ομιλίας. Ο Άρνολτ Χάτς είναι ο επόμενος ομιλητής. Κύριε Μπαρνιέ, επειδή προέρχομαι από τη Βόρεια Ιρλανδία που έζησα πολλά χρόνια τρομοκρατίας, θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν ε, τελωνιακά σύνορα μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Είναι απαρχαιωμένο αυτό το πλαίσιο εμάς μας ταπείνωσε αυτή η συνθήκη γιατί βασιζόμαστε στο 70% του εμπορίου μας ε, με την δημοκρατία της Ιρλανδίας. Γιατί τι θα πρέπει να μην μπορεί να αποφαίνεται και η Εθνική Συνέλευση της Βορείου Ιρλανδίας. Η Συμφωνία Μηχανισμού Ασφαλείας ε, για το backstop θα είναι ολέθρια ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια του ρυθμιζόμενου πλαισίου που θα ισχύσει στο Δινεκές. Θα πρέπει να μας ε, βγάλετε από αυτά τα δεσμά γιατί θα παραμείνουμε μόνιμα φυλακισμένοι. Είναι προς το συμφέρον, όλων αυτό να επιληθεί ειρηνικά. Λάβετε υπόψη τις ευαισθησίες ε, της Βορείου Ιρλανδίας, κύριε Μπαρνιέ. Έντα Ευχαριστώ πολύ. Ζω σε μία κομιτεία στα σύνορα της Ιρλανδίας και ανησυχούμε ιδιαίτερα για το Brexit. Πολλές φορές αναρωτιέμαι κατά πόσο οι υπέρ του Brexit, ε, κατά πόσο γνωρίζουν τι κάνουν στον κοινό, ε, στον κόσμο, στο λαό. Δεν μπορούμε να έχουμε σκληρά σύνορα. Θα ε, πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ασφαλείας. Ως αγορότης ξέρω ότι θα έχουμε ολέθριες συνέπειες στην αγορά. Θα είναι πολύ δύσκολο για μας να πουλούμε και να αγοράσουμε τρόφιμα υψηλής ποιότητας. Δεν καταλαβαίνω πώς οι Βρετανοί μας αφαιρούν αυτές τις δυνατότητες, πώς δεν αφήνουν τους νέους να εργάζονται και να σπουδάζουν σε όλη την Ευρώπη. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα συμβεί στις κοινότητές μας, προσπαθούμε να άρουμε τα προσκόμματα και τώρα τα δημιουργούμε. Πρόκειται για πραγματικές ολέθριες συνέπειες στους λαούς μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπαρνιέ. Συνεχίστε αυτό σας το έργο. Σας χρειαζόμαστε. Δεν θέλουμε να νοδούμε. Να μην ε, υπερβαίνετε το χρόνο σας. Ο κύριος Πασκάλ Μαγκά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Μπαρνιέ. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω το έργο σας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, ε, έτσι ώστε να δούμε ποια θα είναι η έκβαση για να βγούμε κι εμείς αλόβητοι από αυτή τη διαδικασία και πιο δυνατοί. Εγώ ανήκω σε μία περιφέρεια η οποία παράγει κρασί, ένα ε, από τα κρασιά που αγαπούν οι Βρετανοί, τη σαμπάνια. Είναι οι κύριοι εισαγωγής και ίσως και οι πρώτοι καταναλωτές. Κύριε Μπαρνιέ, μπορείτε να μας εγγυηθείτε για το μέλλον, δηλαδή ότι οι Βρετανοί θα μπορούν να πανηγυρίζουν με σαμπάνια και ότι η παραγωγή μας θα μπορούν να εξάγουν σαμπάνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ καλή ερώτηση ο κύριος Έρικ Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και για την εργασία σας. Χαίρομαι γιατί είχα ήδη την ευκαιρία να σας συγχαρώ για την τεράστια αυτή προσπάθεια. Εγώ προέρχομαι από την Ιουτλάνδη, ε, από μια πολύ μικρή πόλη που εξαρτάται από την Αλία. Εσείς μας είχατε επισκεφθεί για να ακούσετε τις ανησυχίες μας, δηλαδή το 40% της αλίας μας γίνεται σε βρετανικά ύδατα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί εσείς εμείνατε στις ε, συμφωνίες αλίας που θα ισχύσουν και στο μέλλον μετά το Brexit. Οι τοπικές αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα ε, και ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές της Βορείου Θάλασσας. Θα θέλουμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα αλίας και στα Βρετανικά ύδατα και θα μπορέσετε να συνεχίσετε προς αυτή την πορεία. David Simons. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι συντηρητικό υπέρ της Ευρώπης από τότε που μπήκα στο συντηρητικό κόμμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε προσωπικό επίπεδο η όλη κατάσταση μου προκαλεί ιδιαίτερη αγανάκτηση. Έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Αναφερθήκατε στην ε, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Δυστυχώ δεν γίνεται όμω κάποια συγκεκριμένη μνήμα ούτε συμφωνία αποχώρηση ούτε στην πολιτική δήλωση. Μολονότι λέτε ότι ε, σε υπουργικό, κοινοβουλευτικό επίπεδο και επίπεδο κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Εμεί, εκπροσωπώντα το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ασχολούμεθα με πολλά πρακτικά προβλήματα προκύπτουν από το Brexit. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την υποστήριξή σα για την συμμετοχή της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης του Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργασία με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ας δώσουμε τώρα τη δυνατότητα στον κύριο Μπαρνιέ να απαντήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι πήραν το λόγο. Ο κύριος Πάης Άντωνη ανέφερε πριν από λίγο τους οικονομικούς και ανθρώπινους δεσμούς. Κοιτάξτε, το λέω για μια ακόμα φορά ότι όλοι λυπούμεθα για την συμφωνία αυτή, αλλά την σεβόμαστε ας μην ξεχνάμε ότι το Μένο Βασίλειο παραμένει μια φιλική χώρα, χώρα σύμμαχος, χώρα εταίρος. Διατηρώντας λοιπόν τις φιλικές αυτές σχέσεις, θα πρέπει με έναν εναλλακτικό τρόπο να παγιώσουμε με διαφορετικό τρόπο, με άλλα νομικά μέσα, αν θέλετε, την οικονομική αυτή εταιρική σχέση που θέλουμε να πετύχουμε, τη συμμαχία στον τομέα της ασφάλειας, καθότι αποφάσισε το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο ότι δεν θέλει πλέον να βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως θα καταβάλω άοκνες προσπάθειες προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτή την φιλόδοξη συνεργασία σε όλους αυτούς τους τομείς που ανέφερα. Κύριε Άντωνη, δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω από αυτά που είπα στον κύριο Μπουκανάν πριν από λίγο. Εγώ δεν μπορώ να παρέμβω στην εσωτερική συζήτηση που γίνεται στο Μένο Βασίλειο για τις ε, σχέσεις, για παράδειγμα, με τη Σκοτία ή την Ουαλία. Υπάρχουν ε, οι αρμόδιοι θύνοντες οι οποίοι διεξάγουν την συζήτηση αυτή. Εμείς ή εγώ τουλάχιστον μπορώ να συζητώ μόνο με την επίσημη και μία κυβέρνηση αυτή του Λονδίνου. Ο κύριος Άντωνη, όπως και ο κύριος Σάμος πριν από λίγο, αναφερθήκατε στο θέμα του συνεχιζόμενου διαλόγου με τις περιφέρειες. Υπενθυμίζω ότι στην πολιτική δήλωση προβλέπεται διαρθρωτική συνεργασία σε υπουργικό, κοινοβουλευτικό, τεχνικό επίπεδο. Πρόκειται για μια συμφωνία βέβαια μεταξύ κρατών μελών και Ηνωμένου Βασιλείου. Ο διαρθρωμένος αυτός διάλογος θα μπορούσε όμως να αφορά και τοπικά και περιφερειακά ζητήματα και, όπως το είπα, μπορεί να ξεκινήσει και ένας θεματικός διάλογος, θα πρέπει να γίνει ο διάλογος αυτός μάλιστα, μετά από δική σας όμως πρωτοβουλία, διάλογος μεταξύ Βρετανικών περιφερειών και Ευρωπαϊκών περιφερειών όσον αφορά τη μελλοντική συνεργασία. Αυτά έχω να σας πω για να σας καθησυχάσω ως προς το ότι θα έχετε σαφώς το μέλλον και τη δυνατότητα να εκφράζεστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ για να ακούει τις ανησυχίες σας. Ο κύριος Χινβόλητα αναφέρθηκε στην ε, επίσκεψη την οποία δεν ξέχασα στη Γιουτλάνδη όπου ασχοληθήκαμε με αλλιευτικά ζητήματα. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ την κατάσταση αυτή για να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη συμφωνία. Δεν μπορεί βέβαια να έχουμε ακριβώ την διασχέση με αυτή που έχουμε τώρα, γιατί αποφάσισαν οι Βρετανοί να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε όμω την δική μας την πρόσβαση στα είδα αλίας καθώς επίσης και την πρόσβαση των Βρετανών στην δική μας την εσωτερική αγορά όσον αφορά τα προϊόντα αλλίας. Ο Πασκάλ Μονζά, όπως και η κυρία Γκαμαρά, ο Κλαβιγιό αναφέρθηκαν στις γεωγραφικές ενδείξεις, υπήρξα και υπουργό Γεωργίας στην Γαλλία και ξέρετε ότι είναι μια χώρα που έχει πολλές γεωγραφικές ενδείξεις, όχι μόνο για τη Σαμπάνια, η συμφωνία λοιπόν στην οποία καταλήξαμε με τους Βρετανούς μας επιτρέπει με τρόπο βιώσιμο να προστατεύσουμε την, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν να κάνουν με τις 3.000 γεωγραφικές ενδείξεις που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ισχύει η προστασία αυτή για όλο το διάστημα αυτό το οποίο θα μεσολαβήσει μέχρι να καταλήξουμε σε μια άλλη συμφωνία για το ζήτημα αυτό. Θα μπορείτε λοιπόν να συνεχίσετε να εξάγετε σαμπάνια στον Ηνωμένο Βασίλειο και εμείς θα μπορούμε να συνεχίσουμε να εισάγουμε ουίσκι σκοτίας. Δύο παραδείγματα δίνω. Κυρία Καμαρά και Λουίς Κλαβιού, προκειμένου να καταφέρει κανείς να φέρει στην εσωτερική αγορά προϊόντα από τρίτη χώρα, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα πρέπει να τηρούνται τα φυτο πρότυπα και όλα τα υπόλοιπα πρότυπα τα οποία επιβάλλουμε για τα προϊόντα τα οποία εισέρχονται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το Γιβραλτάρ αναφερθήκατε στην ε, συμφωνία που επετεύχθη ομόφωνα από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία λέγεται ότι οποιαδήποτε μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να έχει και την σύμφωνη γνώμη της Ισπανίας όσον αφορά το Γιβραλτάρ. Ο κύριος Γκρουπ μας από το Ροτερντάμ, όπως και η συνάδελφό σας από το Αμβούργο, αναφερθήκατε στην προετοιμασία. Πήγα και στις κάτω χώρες και επισκέφθηκα εκεί πέρα το, την τελωνιακή αρχή. 700 νέες θέσεις τελωνιακών έχουμε στις κάτω χώρες, 400 νέες θέσεις τελωνιακών στο Βέλγιο, άλλες τόσες θέσεις ε, στη Γαλλία. Όπως σας είπα, δεν θα έχουμε μια κατάσταση business as usual. Ακόμα και αν έχουμε μηδενικές ποσοστώσεις ή δασμούς, τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν όπως στο παρελθόν. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση όμως θα προκύψουν έλεγχοι, οι οποίοι μπορεί να μην είναι αναγκαστικά δασμολογικοί, αλλά θα είναι έλεγχοι όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων που θα έρχονται πλέον από το Ηνωμένο Βασίλειο, τρίτη χώρα στο μέλλον, προ την εσωτερική αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πάντω για ό,τι κάνετε σε όλε αυτέ τι πιο εκτεθειμένε περιφέρειε για να προστατεύσετε του πολίτε και να προετοιμάσετε τι επιχειρήσει. Κάθε επιχείρηση βέβαια θα πρέπει να προετοιμαστεί με βάση το βαθμό έκθεση που έχει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό αναφέρεται σε αυτέ τι ανακοινώσει τι οποίε έχουμε εκδώσει. Ο Τζέρι Γολφ αναφέρθηκε στην έρευνα, στο πρόγραμμα Εράσμου. Κύριε Γόπα, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία αυτή με έναν άλλον ενδεχόμενο τρόπο. Τη συνεργασία βέβαια την πανεπιστημιακή στα πλαίσια του προγράμματος Εράσμους. Πριν από μερικού μήνε, ε, ε, συναντήθηκα με τον Κιστάφα Ρωσή, γενικό διευθυντή ενό σημαντικού νοσοκομείου στο Παρίσι, ο οποίος ε, ε, διεξάγει έρευνα στον τομέα της ογκολογίας, ο οποίος ε, αναφέρθηκε σε ένα δίκτυο πανεπιστημιακό νοσοκομιακό που έχει δημιουργηθεί για την έρευνα στον τομέα του καρκίνου και μου είπε ότι συνεργάζονται και με το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Ανάλογες πανεπιστημιακές ερευνητικέ συνεργασίες μπορεί να υπάρχουν και για την νόσο του Αλτσχάιμερ ή για άλλε παθήσεις. Προφανώς οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να στοιχιστούν, αλλά απλώ ένα διαφορετικό νομικό ή χρηματοδοτικό πλαίσιο, ακριβώς επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να μην είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κέιτ Φίνι και ο Άρνε Στίνστον αναφέρθηκαν στην Ιρλανδία. Σε καμία περίπτωση δεν ξέχασα την επίσκεψη που έκανα στη Βόρεια Ιρλανδία και έκανα πολλέ επισκέψει στο παρελθόν, στον Τον Κανάν συγκεκριμένα, όπου συνάντησα μια ομάδα γυναικών. Και όντω, κυρία Φίνη, είδα ακριβώ αυτό το οποίο είπατε. Το ζήτημα της Ιρλανδίας δεν έχει να κάνει μόνο με δασμούς, με ελέγχου, με σύνορα, με προϊόντα είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τους άνδρες και τις γυναίκες οι οποίοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η κατάσταση που είχαν δει στο παρελθόν. Θέλουν και επιθυμούν την ειρήνη. Και η ειρήνη οικοδομήθηκε χάρη στο θάρρος ανδρών και γυναικών. Και έχουμε και δύο βραβεία Νόμπελ από την Βόρεια Ιρλανδία που συνεισέφεραν πάρα πολύ στο να παγιωθεί η ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μέσω της προπολογισμού της, μέσω των πολιτικών της πραγματικά πλαισιώνει και στηρίζει την προσπάθεια αυτή για την ειρήνη. Η απάντησή μου λοιπόν είναι σαφώς καταφατική. Οπουδήποτε και να βρεθώ στο μέλλον, οποιοδήποτε πόστο και να αναλάβω, σε κάθε περίπτωση θα προστατεύω, θα προασπίζω τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Και απευθυνόμενο στον κύριο Χάν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για ταπείνωση. Πού έγκυται τελικά η ταπείνωση στην οποία αναφερθήκατε. Καταλήξαμε σε μια συμφωνία αποχώρηση με το Ηνωμένο Βασίλειο στα πλαίσια του που στα πλαίσια του οποίου εκπροσωπείται και η Βόρεια Ιρλανδία, και η οποία είναι αποφελής, θεωρώ, για το σύνολο της Ιρλανδικής νήσου. Και το backstop το οποίο αποδοκιμάσατε Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένα backstop το οποίο το συμφωνήσαμε μαζί με την κυβέρνηση του Μένου Βασιλείου και είπαμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει ίστατη λύση. Θα κάνουμε κάθε τι για να μην το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά πρέπει να υπάρχει στο πλαίσιο συμφωνίας ω εγγύηση. Στον Βασίλειο Όρτα τώρα θα ήθελα να πω ότι Είμαστε έτοιμοι να πραγματευτούμε μια φιλόδοξη συμφωνία στον τομέα του εμπορίου, όπω το επιθυμείτε κι εσεί, λαμβάνοντα υπόψη τι κόκκινε γραμμέ του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώ επίση και τη δική μα την ταυτότητα και τι αρχέ μα. Η μεταβατική περίοδο είτε είναι 21 μήνε ή παραπάνω, θα εξαρτηθεί τελικά από την ίδια την συμφωνία αποχώρηση. Η νομική βάση εκεί βρίσκεται. Πρέπει πρώτα να εγκριθεί αυτή η συμφωνία και μετά θα δούμε πώς θα συμφωνια αποχωρηση η μεταβατική περίοδος. Έχουμε ακόμα πω θα διαμορφωθει η μεταβατικη περιοδο εχουμε ακομα δηλαδή τα καταφέραμε, μένουν εννέα ομιλητές έχουμε διατηρήσει, έχουμε μάλλον κρατήσει τα όρια του χρόνου. Αν μπορεί να μείνει λίγα λεπτά μαζί μας ακόμα ο κύριος Μπαρνιέ. Δίνω το λόγο αμέσως στον συνάδελφο Πρίγκο Εζουέλο. Ευχαριστώ πολύ. Στις 26 Μαΐου, πέρα από τις ευρωεκλογέ θα έχουμε και δημοτικές εκλογές στην Ισπανία υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τους 240.000 Βρετανούς που έχουν απογραφεί και που ζουν στις παράκτιες περιοχές. Είναι 13.000 στη Μούρφια από όπου προέρχομαι και ας μην μιλήσουμε για τους τουρίστες, μιλώ για τους πολίτες, ε, τους Βρετανούς που ζουν στην Ισπανία, πληρώνουν φόρους στην Ισπανία, είναι οι γείτονέ μας, είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας και δεν ξέρουμε κατά πόσο έγκαιρα θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στις ε, δημοτικές εκλογές. Κατά πόσο δηλαδή θα μπορέσουν να είναι και υποψήφοι για τις εκλογές αυτές δεν ξέρουμε τι θα γίνει εάν δεν φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Θα πρέπει να γίνει διμερή συμφωνία με την Ισπανία. Είναι κάτι το πολύ αρνητικό στις διμερείς αυτές σχέσεις. Σας ευχαριστώ. Ντορίν Χουντάρ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπαρνιέ, είχα το προνόμιο να συμμετάσχω στο έργο της Επιτροπής Περιφερειών όλα τα τελευταία χρόνια και εκτιμώ ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο προέβημε σε ανταλλαγή πληροφοριών. Αναπτυχθήκαμε και μαθαίνουμε ημένα από τους ΔΕ. Και ζητώ συγγνώμη από όλες και όλους σας για αυτή την ε, φρικτή ε, πράξη ε, που θα βλάψει και εσάς και εμάς. Όλοι θα υποστούμε την απώλεια την τελευταία τριετία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υφιστάμεθα ε, το βάρος διαρκών ε, καυγάδων, ε, επιχειρημάτων από την άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά, με ψευδείς υποσχέσεις, με ψέματα και βεβαίως τώρα ένα διέξοδο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Εγώ ψήφισα υπέρ της παραμονής. Ε, ζω σε μια πόλη που ψήφισε Remain και σε μια περιφέρεια που παρόλο που έχει χιλιάδες εξαγωγής ψήφισε υπέρ της ε, ε, αποχώρησης. Δεν μπορούμε καν να επανδρώσουμε ε, να στελεχώσουμε επαρκώς τα νοσοκομεία μας χωρίς προσωπικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βοηθήστε μας να ανακόψουμε αυτήν την διαδικασία και να μπορέσουμε να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκατομμύρια από εμά θα σας ευγνωμονούμε. Ο κύριος Έμιλ Μποκ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπαρνιέ, η Βρετανική αποχώρηση είπατε κι εσείς ότι είναι μια αμοιβαία δυσμενής ε, υπόθεση. Δεν έχει νόημα να συζητήσουμε σήμερα για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ. Όμως, ποτέ πια. Αυτό είναι το δίδαγμα. Και πρέπει να δώσουμε περισσότερο, περισσότερη περισσότερο βάρος σε μια ολοκλήρωση ευρωπαϊκή Ένωση εκ των κάτω και όχι εκ των άνω. Δηλαδή να ακούσουμε περισσότερο την φωνή του κόσμου, του, λαού, των πολιτών και όλων των επιπέδων αυτοδιοίκηση. Δεύτερο θέμα. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Βρισκόμαστε μπροστά στο Brexit. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να περιορίσουμε τις ζημιές. Damage control δηλαδή στα αγγλικά. Και είναι θαυμάσια δουλειά που κάνατε κύριε Επίτροπε ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που είναι πράγματι καλύτερη δυνατή. Μια συγκεκριμένη ερώτηση. Εδώ αφορώνται οι ζωές 4,3 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία. Ποια θα είναι η νομική τους κατάσταση εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία. Έχουμε λύση για την περίπτωση που θα υπάρξει συμφωνία. Αν όμως δεν υπάρξει από του χρόνου, τι θα γίνει. Ακολουθεί ο κύριος Λόγκαν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κύριε Μπαρνιέ για το έργο σας. Σημειώνω με πόνο καρδιάς ότι προχωρούμε στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων και είναι γνωστό ότι θα υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις σε πολλές περιφέρειες της Ευρώπης και αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των εθνικισμών. Πρέπει να συνεχίσουμε να εξηγούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να διατηρήσουμε την ενότητά της. Το Brexit δεν σημαίνει το τέλος της συνεργασίας. Πρέπει να σημαίνει την έναρξη μιας νέας φάσης συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχω μια ερώτηση. Ο Γενικός Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δήλωσε προ λίγων ημερών ότι το Ηνωμένο Βασιλείο μπορεί να αποφασίσει μόνο του να μην συνεχίσει το Brexit. Μπορεί να αποφασίσει μονομερό. Ερωτώ λοιπόν, εάν λάβει τέτοια απόφαση το Ηνωμένο Βασίλειο, θα υποδεχτείτε ξανά το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ήδη έχουμε υπογράψει σχετική ε, συμφωνία με την Ουαλία για να διατηρήσουμε ζωντανέ τις ε, συνεργασίες. Ακολουθεί η κυρία Φόρντ. Η Ιρλανδία υφίσταται τις συνέπειες του Brexit. Εκατομμύρια τόνων προϊόντων εξάγονται από το λιμάνι του Κόρκ χωρίς να περνούν από την χερσαία Μεγάλη Βρετανία. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλα τα ενδεχόμενα σενάρια. Το Brexit θα χρειαστεί ιδιαίτερες λύσεις για την ιδιαίτερη γεωγραφική θέση της Ιρλανδίας και τις εμπορικές της ανάγκες. Χρειάζονται προτάσεις για να διατηρηθούν οι σχέσεις και οι μεταφορές μέσω της Βόρειας Θάλασσας και των ε, και τις επαφές με τα γαλλικά λιμάνια. Η γεωγραφία παίζει σημαντικό ρόλο. Η γαλλική οδός είναι σημαντική για να έχουν πρόσβαση τα προϊόντα μας σε Γαλλία, Πορτογαλία και τα ε, άλλα λιμάνια της ε, Μεσογείου. Μπορώ να σας πω λοιπόν κύριε Μπαρνιέ κάτι στα κέλτικα που είναι η γλώσσα των Ιρλανδών. Ευχαριστώ πολύ. Μάργαρετ Λίσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προέρχομαι από μια μικρή πόλη στη βορειοδυτική Αγγλία. Οι περισσότεροι στην πόλη μου ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης. Και όμως προσφέρουμε υπηρεσίες ε, μηχανικών και στην Airbus και στη Rolls Royce. Και εκεί απασχολούνται πολλοί. Η μικρή μας πόλη βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια, εν μέρη και χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσελκύουμε νέες επιχειρήσεις. Το να εγκαταλείψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας αφήσει εμάς στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς φωνή στην Ευρώπη και ούτε καν στην κεντρική μας κυβέρνηση. Φοβούμε λοιπόν για την μου και φοβούμε τι συνέπειες θα έχει η απόφαση για αποχώρηση. Είναι απαράδεκτη η έλλειψη ανεκτικότητας για τις άλλες φωνές. Όποια και αν είναι η έκβαση της ψηφοφορίας στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, η ζημιά έχει γίνει και στο Ηνωμένο και στην Ευρώπη. Εγώ θα συνεχίσω να ελπίζω ότι θα υπάρξει δεύτερο δημοψήφισμα για να ανατραπεί το Brexit. Και ευχαριστώ ε, και εσάς κύριε Παρνιέ που καταβάλατε κάθε δυνατή προσπάθεια υπό δυσχερέστατες συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ. Σαμουήλ Αζοπάγκη. Κύριε Πρόεδρε και εσείς κύριε Παρνιέ προέρχομαι από την Μάλτα με ισχυρές σχέσεις και δεσμούς με το Ενωμένο Βασίλειο και μέλος βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι, επειδή είμαι και δήμαρχος, εξ των Βρετανών που ζουν στην ε, πόλη μου και των πολλών φίλων που έχουμε στο Ενωμένο Βασίλειο, έχω δύο ερωτήσεις προς εσάς. Υπάρχει τρόπος να προστεθούν οι Βρετανοί που θέλουν να παραμείνουν, διότι εν τέλει είναι Ευρωπαίοι πολίτες και τους αφαιρούν τα δικαιώματά τους παρά την θέλησή τους. Υπάρχει οτιδήποτε που μπορεί να γίνει, μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι που παραμένουν, που επιθυμούν να παραμείνουν, ώστε να διορθωθεί η κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ. Δίκλαν Μακδόναλντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ορισμένοι πολιτικοί ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου βάζουν την εξουσία πριν από τους ανθρώπους. Γι' αυτό το Brexit θα έχει ολέθριες συνέπειες όχι μόνο στην παρούσα γενεά, αλλά και στις επερχόμενες αν δεν υπάρξει συμφωνία. Στη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχουν πολιτικοί κατά του backstop και πολλοί commuters μεταβαίνουν τα σύνορα για να δουλέψουν στη μία ή στην άλλη πλευρά της Ιρλανδίας δεν θα πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Στην, σε μία κομιτεία έγινε λόγος για την πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει στον τομέα της, του πολιτισμού και της κληρονομιάς με τη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό ελέγχθη σε μία ε, οργάνωση κομιτιών. Ελπίζω να εστιάσετε όπως συνήθως την προσοχή σας στη στάση των 27 μελών. Ε, Βασισλάφ ε, Τρινκά, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε και σας κύριε Μπαρνιέ, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου σημαίνει ότι 70 έως 80 χιλιάδες Σλοβάκοι πολίτες θα αντιμετωπίσουν σοβαρά γραφειοκρατικά προβλήματα. Πρόκειται κυρίως για πολίτες από την Ανατολική Σλοβακία οι οποίοι εγκατέλειψαν την πατρίδα για να βρουν δουλειά. Μεγάλος αριθμός των πολιτών αυτών αντιμετωπίζει προβλήματα τώρα με, με το νομικό τους καθεστώς. Είναι ασαφές ακόμη, ακόμα και σε περίπτωση soft Brexit, πώς ε, θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή. Θα εξαρτηθεί από την τελική συμφωνία για το Brexit. Όμως για την περιφέρειά μας της Ανατολικής Σλοβακίας η κατάσταση είναι πολύ δυσχερής. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για την έξοδο και καταλήξουμε σε hard Brexit, τότε μετά από τη μεταβατική περίοδο πολλές δεκάδες χιλιάδες Σλοβάκων θα χρειαστεί να επιστρέψουν και είναι σημαντικό η Επιτροπή Περιφερειών να προβλέψει σχετικά μέτρα για να αντιμετωπίσει τις ε, συνέπειες της επιστροφής αυτής. Χρειάζεται λοιπόν να δράσουμε ώστε να υπάρξουν λύσεις και συγκεκριμένα βήματα στην περιφερειακή πολιτική. Παρακαλώ ολοκληρώστε. Εγώ ζητώ η Επιτροπή Περιφερειών να λάβει υπόψη της το ζήτημα αυτό και να ιδρύσει ειδική επιτροπή η οποία θα αναλύσει τις συνέπειες του Brexit και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για συγκεκριμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μπορούν να ληφθούν τα σχετικά μέτρα. Μα πρέπει να ολοκληρώσετε τώρα. Έχετε ε, μιλήσει τον διπλάσιο χρόνο από τους άλλους. Δίνω το λόγο πάλι τώρα στον ε, κύριο Μπαρνιέ για τελευταία φορά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. σύντομη απάντηση στον κύριο Αλόνσο για το τι συμβαίνει με τους Βρετανούς πολίτες, μεγάλος αριθμός άλλωστε, 1,5 εκατομμύριο, οι οποίοι διαβιούν σε κάποια από τις υπόλοιπε χώρες μέλη. Αφής το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει τρίτη χώρα, όπως το θέλησε. Οι Βρετανοί πολίτες δεν θα μπορούν να συμμετέχουν πλέον σε ευρωπαϊκές εκλογές. Λέω, αυτή τη στιγμή θα έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τι ε, ε, κοινοτικέ, δημοτικέ εκλογέ, που ήταν και το περιεχόμενο τη ερωτήσεω σα, αυτό είναι άλλη υπόθεση, διότι κάθε χώρα μέλο, των 27 λοιπόν, διατηρεί την αυτοδύναμη ε, δυνατότητα μέσα στην εθνική του νομοθεσία να προβλέψει διατάξεις που θα επιτρέπουν σε ε, πολίτε τρίτων χωρών να ψηφίζουν στι δημοτικέ εκλογέ. Όμω αυτή την απόφαση δεν λαμβάνεται πλέον στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στο επίπεδο τη κάθε χώρα μέλου. Πάντοτε σε σχέση με του ε, πολίτε αυτού, ο Εμίλ Μπόκ και ο κ. Αζοπάρδη, αλλά και πριν λίγο ο κ. Τρινκάρτ, μίλησαν για του πολίτε αμφωτέρων των πλευρών. Έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία που θεωρώ ότι αυτή ήταν και η προτεραιότητά μα και η προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολλών ενώσεων για να διασφαλιστεί η διαβίωση των 4,3 εκατομμυρίων πολιτών, αλλά και από τις δύο πλευρές. Δεν είναι μόνο οι 90.000 Σλοβάκοι ε, πολίτες, είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί, πολλές δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί και άλλοι. 3,5 εκατομμύρια από τις δικές μας χώρες ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1,3 εκατομμύρια στις υπόλοιπες χώρες. Τα διάφορα δικαιώματά τους, κοινωνικά και άλλα, το καθεστώ τους μέχρι τέλος του 2020, αυτά είναι εγγυημένα. Εάν κυρωθεί και εφαρμοστεί η συνθήκη αποχώρησης και για τα πρόσωπα αυτά και για τις οικογένειές τους και εφόρου ζωής. Νομίζω ότι είναι πολύ θετική η συμφωνία αυτή και βεβαίως αμοιβαία για τους Βρετανούς. Βέβαια θα πρέπει η συμφωνία όντως να κυρωθεί και να εφαρμοστεί. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, κύριε Μποκ, θα χρειαστεί σε αυτόν τον τομέα προτεραιότητας να λάβουμε μέτρα μονομερή από τη δική μας πλευρά. Δεν βρισκόμαστε σε, δεν, δεν εργαζόμαστε υπό αυτό το πνεύμα, δηλαδή να εργαστούμε στη βάση αυτής της υποθέσεως. Προετοιμαζόμαστε βέβαια, αλλά η υπόθεση τη βάση τη οποία εργαζόμαστε είναι να βρούμε λύση τελικώς και συμφωνία για το Brexit. Ήθελα να πω ακόμη στην Ντορίν Ιντάρτ, την οποία παρακολούθησε, παρακολούθησα και συμμερίζομαι τα συναισθήματά της, ότι η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Είναι η εκπεφρασμένη βούληση της πλειοψηφίας του Βρετανικού λαού μέσω δημοψηφίσματος, το οποίο πρόβλεψε η Βρετανική κυβέρνηση για να εγκαταλείψει όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την Τελωνιακή Ένωση και την ενιαία Ώρα. Εδώ υπάρχουν ε, συνέπειε. δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Είναι η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου και τη κυβερνήσεω του. Βεβαίω μετά ακολουθεί η ε, δημοκρατική βρετανική ε, συζήτηση, την οποία σεβόμαστε, αλλά για την ώρα διαπραγματευόμαστε με τη βρετανική κυβέρνηση και έχει ξεκινήσει μια νομική διαδικασία εγκατάλειψη, αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος ε, Λόγκαν μίλησε για τις ε, συνέπειες και νομίζω όπως είπε ο ίδιος και είναι αυτό που τόνισε και ο Εμίλ Μποκ πρέπει να αποδεικνύουμε την αξία της Ευρώπης διαρκώς. Εξακολουθεί το οικοδόμημα που έχουμε φτιάξει όλοι μαζί να είναι έφραστο. Μας ενώνουν αξίες μια κοινότητα μέσω μιας ενιαίας αγοράς που δεν είναι ωστόσο μονάχα μια ζώνη ελευθερών συναλλαγών. Καμιά φορά οι Βρετανοί δυσκολεύονται να το κατανοήσουν αυτό. Με την ενιαία αγορά φτιάξαμε ένα είδο βιοτόπου, ένα οικοσυστήματο δικαιικού προτύπων, προδιαγραφών για κοινά προϊόντα, για κοινά προϊόντα, πρότυπα για προϊόντα δηλαδή, κοινέ διαδικασίε, κοινή εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Και πάνω από όλα αυτά βεβαίω έρχεται μια κοινή δικαιοδοσία, ένα κοινό δικαστήριο. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα, μια απλή ζώνη ελευθερών συναλλαγών. Και γι' αυτό μας σέβονται οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι, διότι αυτή η ενιαία αγορά, ξαναλέω, είναι ένας χώρος κοινή συμβίωση τόσων εκατοντάδων εκατομμυρίων και ε, πολιτών και επιχειρήσεων. Αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ξυλωθεί από τη στιγμή που θα φύγουν οι Βρετανοί, οι οποίοι οφείλουν να σέβονται το ποιοι είμαστε. Όπως και εμείς βεβαίως σεβόμαστε την θέλησή τους να ξαναγίνουν αυτόνομοι. Θα πω στον κύριο Λόγκαν ότι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, πρέπει να αποδεικνύουμε την αξία της Ευρώπης σε κάθε ευκαιρία ώστε να ανταποκριθούμε καλύτερα και στις ανησυχίες των πολιτών. Θα πω επίσης ότι δεν μπορώ να σχολιάσω απόφαση του δικαστηρίου την οποία δεν γνωρίζω και η οποία θα δημοσιευθεί την Δευτέρα στις 9 το πρωί από ό,τι έχει ανακοινώσει ήδη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η κυρία Φόντ μίλησε για τις συνέπειες του Brexit στην Ιρλανδία Σα είπα και ο ίδιος ότι το Brexit δεν προσφέρει απολύτω καμία προστιθέμενη αξία και βλέπει κανεί τα πιο πολλά αρνητικά στην Βόρεια Ιρλανδία διότι ε, προκαλεί πρόβλημα σε μια διαδικασία ειρήνευσης και οδηγεί ενδεχομένως σε μια οπισθοχώρηση. Εμείς είπαμε θα στηρίξουμε την Συμφωνία της Μεγάλης παρασκευή με κάθε τρόπο και ευχαριστώ ιδίω τον Τίσακ, τον ε, Ιρλανδό Πρωθυπουργό και όλη την κυβέρνησή του για το φιλικό κλίμα συνεργασίας το οποίο μας επέτρεψε να φτάσουμε σήμερα εδώ όπου είμαστε. Και θα πω στην κυρία Φόρντ επίσης για τους διαδρόμους σύνδεσης μεταξύ Ιρλανδίας και του υπολείπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα γνωρίζει καλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το τι μπορεί να γίνει σε ό,τι αφορά την διατήρηση των, ε, διαδρόμων αυτών. Και βεβαίως η αρμόδια επίτροπος εργάζεται επ' αυτού. Η Λίσμαν μίλησε για τις συνέπειες για τη Rolls Royce και την αλυσίδα προμηθειών. Δεν θα μιλήσω για εσωτερική βρετανική πολιτική, αλλά οφείλω να πω ότι για τις βρετανικές επιχειρήσεις, και η Rolls Royce είναι από τις μεγαλύτερες, δεν θα είναι πλέον business as usual και σε ό,τι αφορά ιδίω τις, τις αλυσίδες αξίας, διότι η αποχώρησή τους από την ε, ενιαία αγορά θα οδηγήσει καμιά φορά και σε θράψη των αλυσίδων αξίας. Ε, θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Μακδόναλτ στην Ιρλανδία, για την Ιρλανδία αναζητήσαμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα και νομίζω ότι αυτό στο οποίο καταλήξαμε είναι θετικό για την οικονομία του νησιού. Έστω και αν πρέπει κανεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Brexit. Αλλά το ίδιο και για τη Βόρεια Ιρλανδία. Προσπάθησα να απαντήσω σε όλες και όλους και με τη βοήθεια των συνεργατών μου έχω ε, σημειώσει όλε τι ερωτήσει. σα. Η Task Force της οποίας ηγούμε ε, σημειώνει και είναι στη διάθεσή σα να δώσει απαντήσει. Μπορείτε να μα γράψετε και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάθε μία και σε κάθε έναν από εσά. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή Περιφερειών. Cher Monsieur Barnier, vous voyez à la Αγαπητέ κύριε Μπαρνιέ, βλέπετε μόνο και μόνο από το χειροκρότημα αυτό ότι πραγματικά ανταποκριθήκατε στο ύψος των περιστάσεων και πραγματικά σας ευχαριστώ που παραμείνατε μισή ώρα παραπάνω από ό,τι προβλεπότανε. Το εκτιμούμε όλους σε αυτό. Είχαμε, δώσαμε το λόγο σε όλους τους συναδέλφους που τον ζήτησαν. Καλή συνέχεια στο μέλλον. Και σε κάθε περίπτωση με το σημαντικότατο αυτό κείμενο, το ογκώδες κείμενο το οποίο έχει ιστορική σημασία, θα καταφέρουμε να διαμορφώσουμε καλύτερα την ιστορική μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε σχεδόν την ημερήσια διάταξη. Ξέρω ότι ε, δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση όσον αφορά την εκλογή των μελών του Προεδρείου. Έχετε τον κατάλογο ενώπιόν σας. Και έχουμε επίσης ε, και νέα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Στις 6 ε, και 7 Φεβρουαρίου θα γίνει η επόμενη συνοδός μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην οργάνωση της ε, συνόδου αυτής ολομελίας που εμπειρήχε πολλά σημεία στη μερίσια διάταξη. Ο πρόεδρος ευχαριστεί τους διερμηνείς. Εύχομαι σε όλους ε, καλά Χριστούγεννα, καλές διακοπές, ξεκουραστείτε καλά γιατί θα έχουμε ακόμα πολλή δουλειά το 2019 στο τέλος της θητείας μας. Καλά Χριστούγεννα, καλές διακοπές.